Chers collègues, je pense qu'on peut commencer. Επειδή συνάδελφοι, αν δεν απατώμε να αρχίσουμε. Caraïbes, Pacifique et les Émirats Arabes Unis. Suite à la demande. Μετά από αίτημα έγκρισης του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 7 και 218 παράγραφο 6 της συνθήκης η κυρία Γαβριέλα, η εισηγήτριά μας, προετοίμασε την έκθεσή της. Καμία τροπολογία δεν κατατέθηκε και γι' αυτό κυρία Γαβριέλα θέλετε μήπως να λάβετε και το λόγο. Θέλει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ όλους τους κοιόδης για την επικοδομητική μας συνεργασία για τις ανταλλαγές απόψεων και να τονίσω τη δέσμευση του Κοινοβουλίου επ' αυτού του τόσο πολιτικού και συμβολικού εργαλείου που είναι οι θεωρήσεις. Και επιμένω ακόμη μία φορά στην αναγκαιότητα για μας ως Ευρωβουλευτάς να έχουμε μεγαλύτερη πληροφόρηση από την Κομισιόν ως προς την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και επιμένω ότι η υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή πριν την επίσημη επικύρωση του Κοινοβουλίου είναι κάτι με το οποίο δεν συμφωνούμε και πρέπει να το ξαναδούμε την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους ακόμη μια φορά για την εξαιρετική μας συνεργασία. Ευχαριστούμε κυρία Γαβριέλα. Τώρα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Είναι όλοι έτοιμοι με την κάρτα τους. Nous allons voter Θα ψηφίσουμε την κάθε συμφωνία χωριστά. χωριστά. Alors, Euh, pour le premier, pour le Dominique, le vote est ouvert. Η πρώτη για τη Δομινίκα. Άρχεται η ψηφοφορία. Έλξε. Έλξε. Εγκρίνεται. Μετά η Γρενάδα. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Εγκρίνεται. Μετά Αγία Λουκία. Άρχεται. Έληξε. εγκρίνεται. Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες άρχεται. Έληξε. Εγκρίνεται. Τριάς και τον πάγκο άρχεται. Έληξε εγκρίνεται. Σαμόα άρχεται. Έληξε. Εγκρίνεται. Ανατολικό τιμόρ άρχεται. Έληξε. Εγκρίνεται και αυτό. Βανουάτου άρχεται. Έληξε. Εγκρίνεται. Και η τελευταία Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα άρχεται. Έληξε. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Γαβριέλα. Σας υπενθυμίζω συνάδελφοι ότι στην Ολομέλεια θα περάσει το θέμα το Δεκέμβριο. Τώρα το επόμενο σημείο επόμενη ψηφοφορία μάλλον. Τεκμήριο αθωότητος. Άρχεται. Έληξε. Εγκρίνεται. Και προφορική ερώτηση για την Ουγγαρία. Άρχεται. προφορική ερώτηση. Έτσι έλξε. Εγκρίνεται και αυτό. Έλξαν οι ψηφοφορίες. Avant de continuer avec l'ordre du jour. Πριν συνεχίσουμε Λοιπόν λοιπόν, συνάδελφοι, πρέπει να συνεχίσουμε. Και το επόμενο σημείο είναι συνεργασία, στατική συνεργασία για την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητα. Τάκ, τάκ, τάκ. Πρέπει να συνεχίσουμε, είπα, έχουμε και άλλα σημεία στην ημερήσια διάταξη. Το επόμενο θέμα είναι η στρατηγική συνεργασία για την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητα και της τρομοκρατίας μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Ευρωπόου. Η Προεδρία του Συμβουλίου θα υποβάλει σύντομα την εισήγησή της για τα έγκριση των συμπερασμάτων από την Ευρωπόλ τη Συμφωνία και Συνεργασία Διδαμένη των Βαρών Μορφών Εγκληματικότητα με μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και τη Ευρωπόλ. Ο κύριος Βορδέ είναι εδώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε και εσείς, η συμφωνία που μας απασχολεί εδώ είναι καθαρά στρατηγική και αποκλείει αντίθετα από τις κανονικές προσωπικούς χαρακτήρες. Πρόκειται για συνεργασία μεταξύ Ένωσης και Ηνωμένων Αραβικών Ερημινάτων για την καταπολέμηση των βαρών μορφών εγκληματικότητας και τρομοκρατίας. Η στρατηγική αυτή συμφωνία αφορά μόνον ανταλλαγή στρατηγικών πληροφοριών και όχι προσωπικά δεδομένα και προβλέπει την ανταλλαγή εμπειριών, αποτελεσμάτων αναλύσεων και ερευνών για την πρόληψη της οργανωμένης εγκληματικότητας καθώς και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες εκπαιδευτικές. Υπάρχουν μερικοί, μερικές δραστηριότητες εγκληματογόνες όπου μπορούμε να υποφεληθούμε από τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπω απάτε για το φόρο προστιθέμενης αξία και άλλα. Μια αντιπροσωπεία της Ένωσης είχε ήδη πάει στο Αμπουντάμπι, ε, έχει αντιπροσωπεία μόνιμη στο Αμπουντάμπι από το 2013 για μόνιμη συνεργασία με τη χώρα αυτή που είναι σημαντικός εμπορικός μας εταίρος. Για το Συμβούλιο είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν υπόψη ε, τα προβλήματα ασφαλείας επειδή η συμφωνία αυτή αποκλείει την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων, είναι βέβαιο ότι η συνεργασία μας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σε τομείς οικονομικά σημαντικούς για την Ένωση είναι ιδιαίτερη σημασία. Ευχαριστώ. Euh, Κύριε Μπορτέ, ο εκπρόσωπος της Europol θα ήθελε να λάβει το λόγο. Monsieur Neumann, vous avez la parole. Είδε το λόγο. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, συμφωνώ με τη σημασία των συμβουλίων του γιατί πρόκειται για εξαγωγή μη προσωπικών δεδομένων, αλλά είναι στρατηγική ε, ε σημασία και χαρακτήρα. Οπότε, και αυτόν τον τρόπο τώρα ε, είμαι θα θέση να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε την λήψη πληροφοριών σε κάποιους σημαντικούς τομείς όπως η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά επίσης και ε, όσον αφορά τις απάτες αλλά και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Χωρίς αυτή την ε, συμφωνία οι υπηρεσίες μας πληροφοριών δεν θα είχαν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία τώρα μας ε, δίνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οπότε με την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων τότε θα κάνουμε μια επανεκκίνηση άπαξ και έχουμε βέβαια και τη νέα νομική βάση για την Europol όταν αυτή ε, τεθεί σε ισχύ. Οπότε έχουμε αυτή τη στρατηγική συμφωνία που δεν καλύπτει είπαμε προσωπικά δεδομένα. και μιλούμε ότι τώρα αποφεύγουμε καθυστέρηση διαβίωσης δεδομένων κατά δύο ή τρία έτη. ή τρία έτη υπόψη κατά τη συζήτηση. Ευχαριστούμε κύριε Νόημαν, λέει η τρια ετη να ληφθει αυτο υποψη κατα τη συζητηση ευχαριστουμε κυριε νόημα λεει η προεδρος Και τώρα δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Μουσολίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ και επαυξάνω όσα είπε το Συμβούλιο και Europol και όλα αυτά και εγώ τα τονίζω το, το της σημασίας γιατί είπαμε ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά ε, που τώρα σε επίπεδο επιχειρηματικό θα γίνει βέβαια, δεν καλύπτουν τα προσωπικά δεδομένα, γι' αυτό θα πρέπει να ξεχνούμε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι χώρα η οποία μετασχηματίζεται ε, και γίνεται ε, παράδεισος για το οργανωμένο έγκλημα και ε, την τρομοκρατία. Ήδη από το 1978 έχουμε ξεκινήσει προσπάθεια συμφωνίας σε σχέση και με τις άλλες χώρες του κόλπου, αλλά αυτή η συμφωνία αφορούσε ε, οικονομική και τεχνική συνεργασία. Τώρα όμως θέλουμε να προλάβουμε, να καταπολεμήσουμε το, τη σοβαρή εγκληματικότητα και την τρομοκρατία με αυτή τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών ε, και όσον αφορά την ε, μέθοδο πρόληψης τη διαδικασία λήψης των πληροφοριών και στατική ανάλυση. Γνωρίζουμε καλά ότι πρόκειται να ολοκληρωθεί τώρα η αναθεώρηση του κανονισμού ή του καταστατικού της Europol και θα πρέπει επομένως αυτό να μας οδηγήσει σε όσο είναι πιο μεγάλη ευελιξία της Europol. Μια που έρχεται και αυτό να συμπέσει ε, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή τη σύνοψη αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστούμε κύριε Μουσολίνη, κύριε για και τώρα δεν το λόγο στον κύριο Κέρκοπ και κατόπιν κύριε Κάμον. Κέρκοπ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σα πω δύο λόγια. Λόγια συμφωνίας μου με την ε, εισήγηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε το προς τα πού πάει ο κόσμος και τι είδους απειλές διαφαίνονται. Τα Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα βεβαίως αποτελούν τώρα ένα μεγάλο σταυροδρόμι διακίνησης ε, προσώπων ε, πέραν της συμπορικής σημασίας της περιοχής αυτής. Οπότε στα πλαίσια αυτά είναι αναπόφευκτο και εμείς να αναπτύξουμε συνεργασία για σοβαρά έγκλημα και για τρομοκρατία με την χώρα εκείνη. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό βήμα που γίνεται τώρα. Και επίσης σας τονίζω ότι η Δανία, το μέρο Βασίλειο και η Ιρλανδία πρόκειται να προσχωρήσουν σε αυτήν την συμφωνία. Δεν πρόκειται να αυτοεξαιρεθούν δυνάμει των διαφόρων κανόνων και πρωτοκόλων είμαστε αναφανδόν. Υπάρχει και επίσης η Europol μας έχει αποδείξει ότι έχει την εμπειρογνωμοσύνη η οποία τώρα θα ωφελήσει και τα Εμμυράτα μέσω της συμφωνίας. Πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας. Πρόκειται για υψηλά επίπεδα, υψηλά στάνταρ τα οποία μπορούμε τώρα με τις χώρες εταίρους μας να τα εξελίξουμε κι άλλο. Οπότε σημαντική συμφωνία και σημαντικό και το τι θα ακολουθήσει ευκαιρίες για να αντιμετωπίσουμε διάφορες ανησυχίες, διάφορες απειλές που διαχρονικά μας έχουν ταλαιπωρήσει. Άρα αυτά είναι καλά μαντάτα πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ευχαριστούμε κύριε Κέρκο. Κύριε Κόφμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, δεν αμφισβητεί κανείς ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρας για μας. Ε, το εξηγήσαμε ενδελεχώς ε, και είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε με αυτή τη χώρα για την πάταξη της εγκληματικότητας και του, τερο... του Υπάρχει μία ερώτηση που έχει να κάνει με την επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία και με την Βεωσνία Ερζεγοβίνη που θα ε, συζητήσουμε αργότερα. Ε, είναι αυτά τα ζητήματα μέσα στον κανονισμό για την Ευρωπόλ. Εμείς ε, έχουμε το δικαίωμα ακρόασης ως κοινοβούλιο και αργότερα θα γίνει αυτό, θα έχουμε δικαίωμα συναπόφασης γιατί μιλάμε για διεθνείς συμφωνίες με τρίτα κράτη. Και δεν μπορώ να φανταστώ ειλικρινά πώς γίνεται ε, όταν είμαστε τώρα, λίγο πριν τον τριμερή διάλογο και την περάτωσή του για τον νέο κανονισμό για την Ευρωπόλ, να μας αναγκάζουν να κλείσουμε αυτή τη συμφωνία βάσει της παλιάς διαδικασίας που ακόμα ισχύει. Για τη δική μας ομάδα σε χρονικό επίπεδο αυτό ήταν άκερο. Περιμέναμε, θα περιμέναμε να βγει ο καινούριο κανονισμό για την Ευρωπόλ και μετά να γίνει κάτι τέτοιο για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν έχει να κάνει με τη συνεργασία ε, με τα Ηνωμένα Αραβικά ε, ε, Εμμυράτα. Θεωρώ ότι αυτά είναι, αυτή είναι σοβαρή, ε, όπως και αυτή με τη Βοσνία ε, Ερζεγοβίνη. Για μας είναι θέμα αρχής λοιπόν. Και θα ήθελα και η Επιτροπή μας ε, να σκεφτεί πώς θα συμπεριφερθεί και στις δύο συμφωνίες. Ευχαριστούμε κυρία Κάουφμαν. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να λάβουν το λόγο. Όχι. Δεν βλέπω κάποιον. Η κυρία σας είπα στην εισήγησή μου ότι όλοι τελούμε εν επιγνώση του τι έγιναν ε, στην τρεμερή διάλεξη για την τροποποίηση του οργανισμού. αλλά ε, είδαμε τι είπε και ο της Κυροπολό ότι τώρα έχουμε μια συμφωνία η οποία έχει συναυθεί με την ε, Βραζιλία δεν είναι κάποια οποιαδήποτε χώρα είναι με τη Βοσνία Οπότε γι' αυτό και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να χάνουμε χρόνο ακριβώς γιατί αυτή η συμφωνία με την Βοσνία είναι πάρα πολύ σημαντική και γι' αυτό και θα πρέπει να προχωρήσουμε στη σύνοψη της συμφωνίας. Ευχαριστούμε κυρία Μουσολίνη. Σας θυμίζω ότι η ωραία των τροπολογιών είναι λίγη στις 19 Νοεμβρίου το μεσημέρι και οι τροπολογίες πρέπει να κατατεθούν βέβαια στα αγγλικά. Επόμενο σημείο, η επιχειρησιακή στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Βοσνίας, Ερζεγοβίνης και της Ευουροπόλ. Με την ίδια διαδικασία. Πρώτα η Προεδρία του Συμβουλίου θα παρουσιάσει σύντομα τις συστάσεις του Συμβουλίου για το θέμα που σας είπα, επιχειρηματική στρατηγική συνεργασία με τη Βοσνία, Ζεζεκοβίνης και Ευρωπόλ. Ο κύριος Μπουρδέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, εδώ μιλάμε για μία τρίτη φορά το λέμε, επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ Βοσνίας, Ζεζεκοβίνης και της Ευρωπόλ για να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων ε, προσωπικού χαρακτήρα. Για την επιχειρησιακές συμφωνίες με τρίτες χώρες πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι όλα αυτά καθαρά λειτουργικά από τη μία και από την άλλη χωριστά τα προσωπικά δεδομένα όπου προβλέπεται προστασία. Σε αυτή τη φάση θα ήθελα να σας πω κάτι που μου φαίνεται πολύ σημαντικό και για τις δύο αυτές πτυχές. Για το Συμβούλιο καμία από τις δύο αυτές διαστάσεις δεν πρέπει να προέχει της άλλης. Γιατί μια επιχειρηματική συμφωνία δεν θα συναυθεί παρά μόνο εάν πληρούνται και οι δύο όροι. Δηλαδή να υπάρχει λειτουργική ωφέλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό είναι η θέληση του Συμβουλίου, αυτό. Τώρα ας επανέλθω σε ορισμένα από τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά. Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι προνομιακοί εταίροι της Ένωσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Και η Ευρωπόλ απαιτεί συνεργασία με όλες τις χώρες της περιοχής. Μπορεί πολλές περιοχές των Δυτικών Βαλκανίων να είναι κριμινογενείς, αλλά από το 11 υπάρχει συνεργασία με την Μακεδονία, με το 12 με την Αλβανία κλπ. και τη Σερβία. Η συμπερίληψη τώρα της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης θα σημαίνει ότι ολόκληρα τα Δυτικά Βαλκάνια συνεργάζονται. Ορισμένες κριμινογενείς δραστηριότητες είναι ιδιαίτερε στη Βοσνία, Ριζεγοβίνη, δουλεμπόριο, εμπόριο όπλων κλπ. Για μας είναι, είναι προτεραιότητα η καταπολέμηση των δραστηριοτήτων του οργανωμένου κλίματος και προσθέτουμε ότι η Βοσνία ταυτίζεται ως διαμεκατακομιστική οδός μεταναστών, πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα τώρα, και Γύρω από αυτό το φαινόμενο βέβαια κυκλοφορούν και εγκληματικά φαινόμενα όπως το δουλεμπόριο και η παράνομη μετανάστευση. Επίσης σας θυμίζω ότι και για τη μετακίνηση τρομοκαρατών υπάρχει δρόμος από τη Βοσνία Αρζεγοβίνη και γενικότερα από τα Δυτικά Βαλκάνια. Τόσο αυτού η Βοσνία Αρζεγοβίνη είναι υποψήφια ε, υψήφιο της Ένωσης και άρα και, στην Ευρωπόλ. Και θα θέλουμε να ακολουθήσουμε την ίδια στρατηγική που ακολουθήσαμε με τη Σλοβενία και την Κροατία με την επιτυχία που γνωρίζετε. Τώρα, για την προστασία των δεδομένων, όπως σας είχα πει και προηγουμένως, το συμπέρασμα, ε, η κατάληξη μιας επιχειρησιακής συμφωνίας έχει ως όρο την κοινή συμφωνία των δύο συμβαλωμένων. Υπάρχουν 44 σελίδες συμφωνία από το 2013 με την Ευρωπόλ για το σύνολο των ρητρών και διατάξεων που πρέπει να σεβαστεί η Βοσνία ριζεγοβινη Η έκθεση αυτή βασίζεται στην ισχύουσα βοσνιακή αλλά και ερζεγοβινιακή νομοθεσία. Μετά από συνεννοήσεις που έκανε η Ευρωπόλ με τις βοσνιακές και ερζεγοβινιακές αρχές. Οι 28 εκπρόσωποι των χωρών μελών κατέληξε τελικά για την προστασία δεδομένων ότι ήταν αποδεκτή αυτή η συμφωνία και δεν υπάρχει κανένας φραγμός πλέον και εμπόδιο για να αρχίσει τη διαπραγματεύσει της Ευρωπόλ με τη Βοσνία και με την Ερζεγοβίνη. Έτσι το Συμβούλιο διπλά ενέκρινε αυτή την έκθεση και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων με βάση ένα υποπτικό όργανο που αντιπροσωπεύει και τα 28 κράτη-μέλη. Τέλος, αν ακόμα παραμένει κάποια αμφιβολία στο Κοινοβούλιο ως προς τη γνωμοδότηση αυτή, θα θέλαμε να τη μάθουμε αυτή την αμφιβολία. Η συμφωνία αυτή είναι απόλυτη προτεραιότητα λειτουργικά και θα μας ωφελήσει σίγουρα συνεργασία με χώρα εταίρο υποψήφια της Ευρωπαϊκής, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως προς το σεβασμό των προτύπων που ισχύουν παντού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπουρδέ. Τώρα ο εκπρόσωπος της Ευρωπόλου, κύριος Νόημαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κάποια επιπλέον στοιχεία για αυτή την συμφωνία, όπως είπε και ο κύριος Μπουρδέ, οι τομεί τους οποίους περιμέναμε περισσότερη συνεργασία με τη Βοσνία Αρζεγοβίνη και μεγαλύτερη εισρωή και ανταλλαγή πληροφοριών είναι αυτές που είναι οι πιο επίκαιρες η παράνομη μετανάστευση, αντιτρομοκρατικά μέτρα και λαθρεμπόριο. Ότι χωρίς αυτές είναι και χωρίς διαμετακόμισης και προέλευσης. Ακούσαμε λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία αυτή τη συμφωνία προηγήθηκε μια πολύ ε, συγκεκριμένη και αναλυτική εξέταση των λεπτομεριών ε, του θέματος γιατί δεν έγινε μόνο θεωρητική εξέταση αλλά και επιτόπου έλεγχη. Έχουμε και το κοινό εποπτικό ε, σώμα της Ευρωπόλ που αποτελείται από εκπροσώπους των 28 κρατών μελών, τα οποία θεώρησαν ότι βάσει της έκθεσης για την προστασία των δεδομένων στη Βοσνία Ερζεγοβίνη μπορούσαμε να κάνουμε συνδιαπραγμάτευση για την ε, συμφωνία γιατί υπήρχε συμμόρφωση με τα στάνταρ. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη όπως ξέρετε είναι χώρα υποένταξη. Είχαμε παρόμοιες εμπειρίες ε, με την Κροατία. Η συνεργασία λοιπόν με μια τέτοια χώρα βάση μια τέτοια συμφωνίας βοηθά ιδιαίτερα τη χώρα να κάνει όλες τις προσπάθειες που χρειάζονται για να μπορέσει αργότερα να ενταχθεί στις δραστηριότητες της Europol. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Μας βοηθά πολύ και το χρησιμοποιούμε για την ενίσχυση της συνεργασίας. Για να συνοψίσω, να πω ότι ελπίζω ότι θα πάρετε υπόψη σας το γεγονός ότι η προστασία των δεδομένων διασφαλίζει ότι θα γίνεται σεβαστή αυτά τα στοιχεία που θέλουμε από την Ευρωπόλ, ότι αυτή η συμφωνία είναι κάτι που έλειπε από την περιοχή των Δυτικών ε, Βαλκανίων και από άποψη ένταξης της χώρας ε, η Ευρωπόλ θα μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να υποστηρίξει την ένταξη της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ευχαριστούμε τον κύριο ε, Νόημαν. Ο ε, άλλος εισηγητής έχει το λόγο τώρα. Κύριος Φοντάνα, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε και το Συμβούλιο και την Europol για το θέμα αυτό όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα ε, γιατί πάρα πολύ συχνά διαπιστώνεται ε, το ότι είναι σημαντικά τα ψηφίσματα και έτσι βλέπουμε πόσο σημαντικά, πόσο, πόσο, πόσο αποτελεσματική είναι ε, αυτή η συνεργασία ε, αυτό ισχύει πάντοτε με, για κάποιες ε, συνεργασίες, για κάποιες μελέτες με ε, τέτοια κράτη και πάντως γίνεται αντιληπτό ότι η συμφωνία αυτή με τη Βοσνία είναι πολύ σημαντική. Είναι στρατηγική η θέση της χώρας, αλλά βέβαια και πολύ λεπτή και έχουμε από εκεί διάφορες κινήσεις και διαδρομές του διεθνούς εγκλήματος. Πάντως ακριβώς ισχύει αυτό το οποίο είπε προηγουμένως η σοσιαλίστρια συνάδελφος ότι είμαστε λίγο στριμωγμένοι μια που γνωρίζουμε ότι είναι μια συμφωνία πήγε στον τριμερή διάλογο ε, έχουμε την Europol που συμμετέχει και σήμερα οφείλουμε να εγκρίνουμε αυτό το σχέδιο κειμένο χωρίς όμως να καταλαβαίνουμε τι είδους timing είναι αυτό που περιτάνευσε. Γιατί όπως είπαμε και πριν από κάνα μήνα πολύ γρήγορα γίνανε όλα αυτά ε, δηλαδή τη δρομολόγηση αυτού του κανονισμού που ακριβώς σήμερα μας προβληματίζει. Καλά κύριε Βοντάνε, ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Ντίας, Ντεμέρα, που είναι συνεισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να πω στους συναδέλφους ότι ήμουν ο εισηγητής σε σχέση με την απόφαση του Συμβουλίου που αποτελεί τη νομική βάση του, της Europol και τώρα ε, αυτό μετασχηματίστηκε σε κανονισμό και, και καταστατικό για την Europol οπότε καταβάλαμε με τους συναδέλφους των άλλων πολιτικών πτερίγων μεγάλη προσπάθεια και έτσι προχωρήσαμε και κλείσαμε πολιτική συμφωνία για τον ε, κανονισμό της Europol. Και τώρα όσον αφορά την καινούργια και οριστική νομική βάση που καλύπτει την ε, Europol. Έχουμε τώρα ε, δύο τριμερείς διαλόγους, ο ένας πέρασε, ο άλλος έρχεται την επόμενη εβδομάδα και αυτό το οποίο για μένα παραλήφθηκε να μνημονευτεί αφορά τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Γιατί εκεί μιλούσαμε για στρατηγική συνεργασία. Και δεν συμφωνώ. Μπορώ να μην συμφωνήσω. Ε, βέβαια και συμφωνώ. Μια που πρόκειται για κάποια θέματα στρατηγικής σημασίας. Ε, επίσης, θεωρώ ότι είναι κάτι το καλό και κάτι το αναγκαστικό το να συνάπτουμε ε, τη συμφωνία με Βοσνία και Ερτζεγοβίνη και πρέπει να σας ενημερώσω συνάδελφοι ότι τη σήμερα ημέρα η Europol έχει συνάψει συμφωνίες στρατηγικού χαρακτήρα με τη Βοσνία, με τη Ρωσία, την Τουρκία και την Ουκρανία. Και έχει επιχειρησιακές συμφωνίες σήμερα με Αλβανία, Αυστραλία, Καναδά Κολομβία, Μακεδονία, Ισλανδία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Ελβετία, ε, Μονακό ε, και είπα αυτό που τώρα προτείνεται τι είναι μια επιχειρησιακή συνεργασία και συμφωνία γιατί το Συμβούλιο θεώρησε ότι πρέπει να εγκρίνει μέσω του Δυτικού Συμβουλίου της Europol τη σχετική απόφαση, ούτω ώστε να έχουμε μια συμφωνία για ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων. Σε αυτό αναφέρθηκε και το Συμβούλιο και η Europol. Αλλά κατά τη γνώμη μου εδώ έχουν άλλους τα πράγματα. Γιατί. Είναι αδιάφορο για ποιο λόγο εδώ υπάρχει αυτή η διάκριση. Γιατί αν συνεχίσουμε την πορεία αυτή που θέλει το Συμβούλιο και η Europol, τότε η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου είναι απλώς μία γνωμοδότηση, μία έκφραση γνώμης. Εγώ όμως ως εισηγητής άλλο πράγμα θέλω και το θέλω για να μην διαταράξω αυτή τη συνένεση που υπήρξε με τη Euro, για τη Europol με τα άλλα πολιτικά κόμματα. Θέλω αυτό και αυτό το θέλουν και τα άλλα πολιτικά κόμματα που συνεργάστηκαν μαζί μου. Είναι δηλαδή ότι όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την ανταλλαγή των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή λειτουργικέ και επίξιακέ συμφωνίε να είναι κάτι το οποίο να διέπεται από τη συναπόφαση. Δηλαδή να συναποφασίζει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Γιατί αν συνεχίσουμε τη σημερινή ρότα, τότε αποκλείουμε το Κοινοβούλιο από τη λήψη αποφάσεων. Οπότε και θα απλώς θα γνωμοδοτεί το Κοινοβούλιο. Πάντως, σε σχέση... Ε, βάσει της αλφάς 934 για την ε, Βοσνία όσον αφορά την ανταλλαγή των δεδομένων έχουμε αυτή τη συμφωνία επιχειρησιακή στρατηγική και αφορά ανταλλαγή των προσωπικών δεδομένων. Δεν μπορεί είναι δυνατόν κανείς να αποφύγει το να φυγούν τα προσωπικά δεδομένα, να μην συζητηθούν. Χρειάζεται επομένω μια απόφαση θετική της ε, ρυθμιστικής αρχής, της ελληνικής αρχής. Ο πάντως εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να γίνει είναι κάτι το οποίο καλύπτει αυτή την ελεγκτική αρχή. Δηλαδή την θέλουμε την τελευταία λέξη να την έχει η Ευρωπαϊκή Εποπτική Υπηρεσία Ελέγχου Προσωπικών Δεδομένων και όχι η, η Europol. Και οπότε, στις 13 Μαΐου του 2015 ξεκίνησε αυτή η διαδρομή, προχώρησε στο Κοινοβούλιο με την διαδικασία της διαβούλευσης. Είπαμε, οπότε παρουσίασε τις προτάσεις στο Συμβούλιο, παρουσία της Europol και η προθεσμία κατάσταση τροπολογιών γνωρίζετε ότι είναι 19η Νοεμβρίου. Και συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριο Φοντάνα. Είναι λογικά. Και λέγω τούτο. Ο κανονισμό για την Europol το Δεκέμβριο τον Ιανουάριο πρέπει να εγκριθεί με συμφωνία πολιτική. Οπότε και έχουμε έτσι πράσινο φως για αυτή την επιχειρησιακή συνεργασία. Οπότε και θα πρότεινα να περιμένουμε την έγκριση του κανονισμού. Πριν από ένα χρόνο κυρία Πρόεδρε με αυτό τελειώνω, έμαθα ότι υπάρχει και άλλη παρόμοια έκθεση που αφορά Βραζιλία, Μεξικό, Γεωργία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και επειδή θέλαμε να δώσουμε περισσότερο πρωταγωνισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι τότε η συνεργασία, δώσαμε 42 ψήφου κατά και 0 υπέρ εκείνη τη συμφωνία. 0-42 ήταν το σκορ. Λάβετε το αυτό υπόψη. Ναι, να συνεργαστούμε με τη Βοσνία. Όμως η συνεργασία να γίνεται δυνάμει της νομικής βάσης όχι απόφαση συμβουλίου αλλά κανονισμού. Κύριε Ντεμέρα, ευχαριστούμε. Πριν συνεχίσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, και πριν δώσουμε σε του ανθρώπου το λόγο, επιτρέψατε μου να ευχηθούμε καλώ όρισαν κάποιοι επισκέπτε από την Σουηδία, για του οποίου έχει προσκαλέσει η κυρία Κοράτσα Μπίλ. Σήμερα θα διαπιστώσουμε πώ δουλεύουμε εδώ στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Καλώ ορίσατε. Τώρα συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Η κυρία Κάφμαν θέλετε το λόγο ή όχι. Πολύ σύντομα νομίζω ότι εμείς ως κοινοβούλιο πρέπει να σκεφτούμε ακριβώς πώς θα συμπεριφερθούμε σε σχέση με τις ε, συμφωνίες που είναι διαφορετικής φύσεως. Ε, είπε ο συνάδελφος ήδη ότι οι διαπραγματεύσεις της Ευρωπόλ πρέπει να κλείσουν ε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Βέβαια θα έχουμε, έχουμε μια άλλη νομική βάση και θεωρώ ήδη ότι εμείς στο Κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίσουμε βάση αυτής της νέας βάσης γιατί είναι διεθνή συμφωνία και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το δικαίωμα συναπόφασης. Και αυτό το δικαίωμα δεν το χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα από το γεγονός ότι και οι δύο συμφωνίες ασχολούνται με διαφορετικά ζητήματα. Ευχαριστούμε κυρία Κάουφμαν. Ευχαριστώ πολύ επειδή είχα εξετάσει και εγώ μια ανάλογη πρέπει να σας πω ότι οι τριμερείς διάλογοι συνεχίζονται πολύ, με πολύ μεγάλη ταχύτητα και ελπίζουμε να είναι έτοιμο το πλήρες έγγραφο όπως γίνεται και με τον τριμερή διάλογο για την Ευρωπόλ. Άρα, άρα είναι πολύ πιθανό να υπάρξει ευτυχής κατάληξη. Κάθε χώρα που δέχεται τέτοια συνεργασία πρέπει να αποδεικνύει ότι εφαρμόζει τα πρότυπα. Και με μεγάλη χαρά άκουσα τα νέα για τη Βοσνία αλλά και για την Ερζεγοβίνη ότι τέτοιου είδους έρευνα έχει ήδη γίνει. Επίσης όμως θα ήταν σημαντικό να δούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες τα αποτελέσματα της έρευνας. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς ποια πρότυπα εφαρμόζονται και να πιστούμε. Και όταν θα γίνει αυτό, δεδομένης και της δύσκολης κατάστασης στα Δυτικά Βαρκάνια, τότε μπορεί να εγκριθεί ένα ψήφισμα και όχι πριν, γιατί τότε θα έχουμε εμπιστοσύνη. Confidence, we have to listen. Γιατί χωρίς εμπιστοσύνη δεν γίνεται. Εμείς χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος για τις τροπολογίες λοιπόν. Πρέπει να δούμε και άλλα έγγραφα και μετά να αποφασίσουμε για την έγκριση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Φαντενάης, θέλετε το λόγο. Κύριε Φαντάνα. Όχι, θέλω να σας πω ότι συμφωνώ με τους αδέλφους, λέει ο κύριος Φοντάνα, και ε, θα πρέπει ακριβώς να δούμε πόσο σημαντικό είναι, αυτό το σύμφωνο. Όχι κάθε αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, μπορούμε έτσι να έχουμε ε, κάποιο νομοθετικό όργανο ε, για τα προσωπικά δεδομένα. Και όταν υπάρχουν αποκλίνουσε απόψει, τότε αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε προτεραιότητα σε ό,τι ενδιαφέρει το Κοινοβούλιο. Που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάτι το τόσο σημαντικό και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Λαδεστίν. δεσμεύεται η γραμματεία μας να δώσει σε όλους τους συναδέλφους τα έγγραφα στα οποία αναφερθήκατε. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία κατά τροπολογιών είναι η 19η Νοεμβρίου. <clears throat> Τώρα πάμε στο επόμενο σημείο που είναι το υπαριθμό 22 πρόσβαση του κοινού ή στα έγγραφα άρθρο 116 που αφορά την περίοδο 2014-2015. Πρόκειται για κάτι το οποίο αφορά την διαφάνεια συγκεκριμένα το θεμελιώδες δικαίωμα της πρόσβασης ή στα έγγραφα κάτι το οποίο κατοχυρώνεται από τον χάρτη δικαιωμάτων της Ένωση το προβλέπετε αυτό ο κανονισμός 1049 και προετοιπομένως στην έκθεση να προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτή την περίοδο 14-15 αλλά τώρα να δώσουμε τον λόγο εις την εισηγήτριά μα την κυρία Φεράρα θα μας παρουσιάσει το σχέδιο κειμένου της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε κυρία Φεράρα. Παρά τα όσα προβλέπονται από τα θεσμικά όργανα, όλα πρέπει πολύ αφηρημένα, μακριά από τους πολίτες που δεν ξέρουν τι γίνεται, που είναι κάτι που δεν ανακατεύεται με τη ζωή τους, οπότε ε, είχαμε την εβδομάδα αυτή, την πράσινη εβδομάδα και περισσότεροι δουλέψαμε στο χωριά και στις πόλεις μας και είδαμε τι λένε οι πολίτες που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στις ε, πληροφορίες αλλά ακόμα και οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να έχουν προσβασιμότητα στην έγγραφα αυτά για να τους ε, ενημερώσουν ε, οπότε κατά κάποιο τρόπο είναι στριμωγμένοι οι πολίτες δεν μπορούν να μάθουν τα δικαιώματά τους τα οποία απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο και αυτό αφορά τον ε, κανονισμό 1049 του 2001, το προβλέπουν και οι συνθήκες και έχουμε το άρθρο 15 του Χάρτη Δημοκρατία Δημοκράτων και έχουμε το άρθρο 11 επίσης για την ε, συνθήκη για την λειτουργία της Βουλής και την συμμετοχική δημοκρατία προβλέπονται ότι επίσης ε, έτσι θα πρέπει τα θεσμικά όργανα να δημοσιοποιούν αυτό το οποίο χρειάζεται ώστε να μπορούν να ξέρουν τι γίνεται οι πολίτες, να υπάρχει ανοιχτός διάλογος, διαφάνεια ε, και αυτό να γίνεται σε τακτικά διαστήματα με γίνεται των πολιτών. Υπάρχει επομένως ακόμα πολλής δρόμος να κάνουμε για να ε, εφαρμόσουμε αυτό που προβλέπει το άρθρο 11 της συνθήκης. Θα πρέπει να καταλάβει ο Ευρωπαίος τι κάνουν ε, αυτοί που εκλέγει, τι κάνουν οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων και τελικά οι πολίτες είναι οι τελικοί κριτές των όσων κάνουμε εδώ και επομένως ε, δεν θα πρέπει να αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μια ένωση γραφειοκρατών. Θα πρέπει να μπορεί ο κόσμος να καταλάβει και να εκτιμήσει αυτά τα οποία κάνουν οι εκπρόσωποι του στα θεσμικά όργανα. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται αυθεντική διαφάνεια αυτό το υπαγορεύει η ίδια η δημοκρατία και η διαδικασία λήψης απόφαση. Άρα πρέπει να κάνουμε εδώ μια επανεκκίνηση, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Και γι' αυτό το λόγο στην έκθεσή μου ετώνησα το πόσο σημαντική είναι η διαφάνεια, η πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων. Αυτό, αυτό θα πρέπει να είναι ο κανόνας και η εξαίρεση να είναι ε, η, η εμπιστευτικότητα όπως ε, λέει ο κανονισμός 1049 ε, και το έχει πει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οπότε ακριβώς που δεν έχουμε μια διοργανική πολιτική που να καλύπτει τον πολίτη και να εφαρμόζει διαφάνεια στην επικοινωνία και μια άμεση δημοκρατία. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς η καθημερινή πρακτική θα έχει διαφάνεια, θα ενημερώνονται οι πολίτες για τα όσα κάνουμε. Τι γίνεται επίση και στο Συμβούλιο. Εκεί βέβαια δεν είναι δημόσιες οι Θα έπρεπε όμως και οι περισσότερες συζητήσεις γίνονται και κλεισμένων θυρών και δεν υπάρχει κανένα έγγραφο, καμία ενημέρωση σχετικά ούτε πριν ούτε μετά αυτές τις συνεδριάσεις. Επίσης όσον αφορά τους τριμερείς διαλόγους αυτές τις διαπραγματεύσει μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και αυτοί οι τρίλογοι, οι τριμμένες διάλογοι γίνονται και κλεισμένων, δεν υπάρχει ούτε μετάδοση στο ίντερνετ, ούτε κανένας είδους δημόσιο έγγραφο, αλλά μετά την τρίτη ανάγνωση έχουμε καταντήσει έτσι να είναι η πάγια πρακτική. Και τελικά έτσι ωφελούνται τα λόμπι και διευκολύνονται και μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Τώρα όσον αφορά του λομπίστες έχουμε κάποια πρόταση στην έκθεσή μας και λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα υποχρεωτικό διοργανικό μητρό των εκπροσώπων των ε, διαφόρων συμφερόντων που δουλεύουν στα θεσμικά όργανα. Και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να δημοσιεύουν όλες αυτές τις ε, πληροφορίες για τις επαφές με τους λομπίστες ε, για τους, ε, τους, τους τι κάνουν οι υπάλληλοι που τους συναντούν οι βουλευτές όλοι τέλο πάντων και στο Συμβούλιο και εδώ και σε σχέση επίσης με κάποιες διεθνείς συμφωνίες που δεν διακρίνονται από υποχρεωτικότητα θα πρέπει και εδώ να δούμε τι θα γίνει και να έχουμε δημοσίευση της διαπραγματευτικής εντολής που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τη λαμβάνει να δούμε επίσης τι γίνεται και με τις διαδικασίες επί παραβιάση του δικαίου και αυτά να είναι δημοσιοποιημένα και να ξέρει ο κόσμος ακριβώς που ήμαρτεν η κυβέρνησή του. Επίσης, όσον αφορά την διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων και εκεί χρειάζεται να υπάρχει διαφάνεια για τις επαφές επιτροπής περιφερειών και κρατών για τα λειτουργικά προγράμματα, τα περιφερειακά κλπ και σας επαναλαμβάνω ότι θεωρώ πως θα πρέπει να εγγυηθούμε περισσότερη διαφάνεια και προσβασιμότητα εις της πληροφορίας και έτσι να επιτρέψουμε στον κόσμο που να μπορεί να έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να κατανοήσει καλύτερα την δυναμική, τη λειτουργία και κυρίως ο κόσμος να έχει επίγνωση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από το κοινωτικό δίκαιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα δίνω το λόγο στους σκιώδεις. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες έχουν σκιώδεις, αλλά μόνο δύο βλέπω στην αίθουσα. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Κοράτσα Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ πλήρως ότι έχουμε μια κοινή πρόκληση να συνδέσουμε τους ε, πολίτες να γίνουν πιο ε, διαφανείς οι διαδικασίες, η λογοδοσία, ο τρόπος ε, που νομοθετούμε, που ε, δαπανούμε το δημόσιο χρήμα, όλα αυτά που πρέπει να γίνουν και υπάρχουν και άλλα τόσα μέχρι να κλείσει αυτό το χάσμα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα λοιπόν τα οποία τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να κάνουν ακόμα περισσότερο, ειδικά το Συμβούλιο. Η Κομισιόν έχει κάνει κάποια πρόοδο. Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο είναι μακράν το πιο διαφανές και ανοιχτό Κοινοβούλιο στον κόσμο με την ε, live αναμετάδοση στο διαδίκτυο όλων των συνεδριάσεών μας για τους ε, πολίτες της Ευρώπης, για τους τριμερείς διαλόγους. Να πούμε καταρχάς τι είναι. Είναι ένας τρόπος διαπραγμάτευσης, ο οποίος ενισχύει και επιταχύνει την λήψη αποφάσεων και την συμφωνία μεταξύ των δύο νομοθετών ε, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τη συνδιαλλαγή η οποία διαρκεί πάρα πολύ. Όλα βέβαια εξαρτώνται και από τον εισηγητή αλλά και από το θέμα. Πρέπει να ε, δώσει λόγο στην Υπόεθνη Επιτροπή, στον, ε, στους σκιώδεις από την κάθε πολιτική ομάδα. Δεν είμαι σίγουρη αν οι πολίτες τελικά θα έχουν κάποιο όφελος από το να συμμετέχουν σε αυτές ε, τις διαπραγματεύσεις γιατί χρειάζεται πραγματικά ένα κλίμα εμπιστοσύνη για να μπορεί κανείς να φτάσει σε συμβιβασμό σε περίπλοκες καταστάσεις. Πολλές φορές είναι ακόμα και αντιπαραγωγικό. Οι πολίτες θέλουν μια νομοθετική διαδικασία, δημοκρατική διαδικασία η οποία θα φέρνει γρήγορα αποτελέσματα με δημοκρατικό τρόπο. Για να μπορέσουμε λοιπόν να κλείσουμε αυτό το χάσμα της δημοκρατίας πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, να αφήνουμε χώρο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, της προσωπικής ζωής, ε, της προσωπικής ακεραιότητας, Όλα αυτά πρέπει να γίνονται σεβαστά. Ακόμα και μια χώρα όπως η Σουηδία που είναι μακράν στο, στην πρώτη θέση όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής του, ε, της διαφάνειας ε, ε, θα πρέπει να γίνουν και εκεί πράγματα. Γενικά, ε, ακόμα και σε μια τέτοια χώρα ε, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διαβάθμισης των εγγράφων. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια ανοιχτή δημόσια συζήτηση με τη συμμετοχή των πολιτών να γνωρίζουν ε, τι διακυβεύεται, ποιο είναι το αποτέλεσμα, αλλά δεν νομίζω ότι το κάθε στάδιο της διαπραγμάτευσης πρέπει να δημοσιοποιείται, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει εμπιστοσύνη κατά τη διάρκεια της ε, διαπραγμάτευσης και εμπιστευτικότητα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα καθ' όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης παρόλα αυτά. Επίσης είναι η ώρα πλέον να κάτσουν τα τρία θεσμικά όργανα και να σπάσουν το διέξοδο για τη δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα. Είναι σκάνδαλο που μπλοκάρεται στο Συμβούλιο εδώ και χρόνια. Το ΕΛΚ θα συνεχίσει να δεσμεύεται και για την λογοδοσία και για την διαφάνεια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Μπίλτ. Ε, επόμενη σκιώδης. Η κυρία Χέτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το σχέδιο έκθεσης ε, το οποίο πραγματικά είναι ένα ντοκουμέντο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, διότι οι πολίτες μπορούν να είναι δραστήριοι, να λάβουν μέρος στη διαδικασία αποφάσεων και στην ουσία εμείς ως αιρετοί ε, μπορούμε να εκπροσωπήσουμε τους εκλογείς μας. Στα κράτη-μέλη λοιπόν και εκτός αυτών ε, εκεί Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε λίγο και να σκεφτούμε τι ακριβώς θέλουμε, γιατί και στα κράτη-μέλη γίνονται αντίστοιχε διαδικασίες. Θέλουμε να μην ε, αλλάξουν τα πράγματα ώστε στο μέλλον να γίνεται πιο δύσκολη η πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα. Μπορεί να μπλοκάρεται κάτι στο Συμβούλιο, αλλά γενικά φαίνεται ότι οι κυβερνήσεις θέλουν να ε, περιορίσουν τη διαφάνεια, το να είναι ανοιχτά τα έγγραφα. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες, κάποια συγκεκριμένα σημεία, ας πούμε στο σημείο 5 λέει ότι τα θεσμικά όργανα δεν είναι ακριβά, ακριβώς όσο ε, προμηθεί θα έπρεπε για να μπορέσουν να βελτιώσουν αυτή τη διαδικασία. Το Κοινοβούλιο λοιπόν προσπαθεί ε, με τον έναν τρόπο και τον άλλον να κάνει τα, πρόγρα... τα έγγραφα δημόσια, ίσως με λάθος τρόπο ακόμα και στα κοινωνικά δίκτυα. Επίσης υπάρχει μια κριτική σε κάποιο άλλο σημείο σχετικά με τους τριμερείς διαλόγους. Οι τριμερείς διάλογοι είναι σημαντικοί από πρακτική άποψη, αλλά πρέπει να είναι όσο πιο διαφανής γίνεται. Ευχαριστώ για το σχέδιο. Χαίρομαι για την καλή συνεργασία με τις συνεργατές με την ε, συντάκτρια και με τους σκιώδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Χέντ. Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει να λάβει το λόγο? Όχι. Σας θυμίζω ότι η κατάθεση των τροπολογιών έχει προθεσμία στις 27 Νοεμβρίου, στις 2. Τώρα αγαπητοί συνάδελφοι να σταματήσω για λίγο, για 30 λεπτά συγκεκριμένα, γιατί Περιμένουμε την κυρία Ρεϊνάλ και τον κύριο Λεπρέχτ που είναι συγκεκριτής για το επόμενο θέμα. Επανερχόμαστε σε 30 λεπτά. Des, euh, des points de l'ordre du jour, par exemple, parce que Madame Plouz, qui était là,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

Chers collègues, je pense qu'on doit commencer déjà notre travail. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τι εργασίε μα Το επόμενο θέμα, το σημείο 23, έχει να κάνει με την, με την υπόθεση σε 362-14 Maximilian Sherms ε, κατά του Data Protection Commissioner. Σήμερα έχουμε τη συνεργάτηδα ε, για το άρθρο 29 που θα μας μιλήσει για το θέμα αυτό. Θα την περιμένουμε. Η οποία αντικαθιστά η κυρία Ρεϊνάλ, την κυρία Μεροτάνο, η οποία έπρεπε να δεν μπόρεσε να, πάει, να έρθει σήμερα στις Βρυξέλλες ε, λόγω έκτακτων ε, γεγονότων από την Γαλλική Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων η κυρία Ρεϊνάλ εργάζεται σε αυτή την ομάδα, όπου είναι υπεύθυνη για τα διεθνή και ευρωπαϊκά ζητήματα. Το ίδιο και η κυρία Πιροτάν είναι η πρόεδρος της ομάδας 29. Είναι συνεισηγήτρια της ομάδας 29 ε, για τις επιπτώσεις του ζητήματος αυτού, της υπόθεσης ΣΕΡΜΣ. Υπάρχει λοιπόν μια θέση της ομάδας εργασίας μετά από την ε, απόφαση του δικαστηρίου και της αρχής για τη μεταβίβαση των δεδομένων. Μετά από αυτό λοιπόν οι συγητές ε, για την προστασία των δεδομένων θα πάρουν το λόγο και μετά οι συνάδελφοι από την Κομισιόν που δεν είναι εδώ αλλά ίσως θα έρθουν αργότερα. κυρία Ρεϊνάλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, καταρχάς παρακαλώ να με συγχωρήσετε γιατί δεν μπόρεσε να προσέλθει η κυρία Ρεϊνάλη ίδια. Θα ήθελε αλλά για λόγους βεβαρημένων εργασ... Ε, του εργασίας δεν μπόρεσε. Μιλάμε λοιπόν για τις επιπτώσεις της απόφασης αυτής του δικαστηρίου για τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων της Εθνικής Αρχής. Καταρχήν, οι ευρωπαϊκές αρχές αποφάσισαν να λάβουν ό,τι με χρειάζεται για να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Είναι βέβαια σοκαριστικό αυτό. Αλλά δεν ήταν και καμία έκπληξη. Και συνεχώς επανελάμβαναν από το 2013 ότι η μαζική επιτήρηση και εποπτεία, η μυστική δεν συμβαδίζει με τις βασικές αρχές της Ευρώπης και είναι απαράδεκτη σε μια δημοκρατική κοινωνία. Δημοσιεύσαμε δύο τεχνικές νομοδοτήσεις το 2014 για αυτό το θέμα και μια πιο πολιτική δήλωση το Δεκέμβριο του 2014. Και εκτός αυτών, από το 2000 έχουμε εκφραστεί για τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν στο εργαλείο αυτό. Ιδιαίτερα μία επιστολή του Φεβρουαρίου 15 προς την κυρία Γιώργα. Επίσης επανειλημμένως είπαμε ότι η λύση για την πρόσβαση ξένων αρχών σε δεδομένα που προστατεύονται από την Ευρώπη εξαρτώνται από διεθνείς συμφωνίες αλλά όχι από συμβατικές υποχρεώσεις σε ιδιωτικά συμβόλαια ακόμη κι αν, αφορούν κοινοτικά όργανα και δεν μπορούν να συγκριθούν με την νομοθεσία των τρίτων χωρών. Τέτοιου είδους εργαλεία θα δημιουργήσουν λοιπόν διαμάχες προτύπων αλλά δεν θα τις λύσουν δεν είναι ο στόχος τους αυτός. Και γι' αυτόν τον λόγο Ζεβετνάφ 29 εκφράστηκε στις 16 Οκτωβρίου πριν από λίγο μετά την απόφαση ζητώντας από τις κυβερνήσεις και τους θεσμούς και των δύο πλευρών του Ατλαντικού μέσα σε τρεις μήνες μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να βρουν μια λύση. Λύση πολιτική, νομική ή τεχνική, ώστε στις Ηνωμένε Πολιτείες να υπάρξει μία ουσιώδης προστασία ισοδύναμη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ιδεοδός θα χρειαζόταν εδώ διακυβερνητική συμφωνία γιατί οι συμβατικές λύσεις δεν αρκούν για να λυθεί τέτοιο πρόβλημα της μαζικής επιτήρησης σε τρίτη χώρα. Μας φαίνεται λοιπόν ουσιώδες αν φανεί ότι η νομική τάξη των Ηνωμένων Πολιτειών δεν συμβαδίζει με του Ευρωπαίου δικαστή τότε ένα νέο σεφάρμπορ, το σεφάρμπορ 2 δεν θα έφερνε μια ουσιαστική λύση παρά μόνο εάν οι εγγυήσει του είχαν δεσμευτικό χαρακτήρα για το αμερικανικό δίκαιο όχι μόνο επί των επιχειρήσεων όπως γίνεται τώρα αλλά και των υπολείπων οργάνων Αναμένοντας λοιπόν την κατάληξη αυτών των διαπραγματεύσεων που ελπίζουμε να έχουν οριζόντιο αποτέλεσμα. Το γάμα 29 θέλησε να επιδείξει κάποιο ρεαλισμό. Καταρχάς, βλέπει ότι το Σέφαρ δεν υπάρχει πια. και άρα οι μεταφορές που γίνονται στα πλαίσια του είναι παράνομες. Αυτή τη στιγμή οι αρχές προσαρμόζουν τα ερωτηματολόγια και τα έγγραφα που απαιτούν για να συμφωνεί με την απόφαση αυτή. Επίσης, με συντονισμένο τρόπο γίνεται καμπάνια ευαισθητοποίησης γιατί φαντάζεστε ότι οι επιχειρήσεις που μεταφέρουν δεδομένα αλλά και οι πολίτες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα. Εξάλλου το 29 θέλησε να εξετάσει και τα υπόλοιπα εργαλεία μεταφοράς δεδομένων. Αποφασίζοντας οι επιχειρήσεις να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία όσο διαρκεί η ανάλυση γιατί δεν μας φαίνεται ρεαλιστικό να αποφασίσουμε ξαφνικά να σταματήσουν όλες οι μεταφορές δεδομένων προς τις Ηνωμένε Πολιτείες αν δεν έχει γίνει πρώτα μία ολοκληρωμένη μελέτη ιδίω ως προς τις εξαιρέσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία και που μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές αρχές. Γι' αυτόν τον λόγο αποφασίσαμε να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος τρίμηνη μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 16 κατά την οποία οι επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία. Μέχρι τότε λοιπόν τι προβλέπει το G29. προβλέπει, α όχι πριν να σας πω τι προβλέπει. Μία υπενθύμηση για τις δικαιοδοσίες που έχουν σήμερα ορισμένες αρχές έχουν δικαίωμα ελέγχου απριόρι. Απαιτούνται δηλαδή άδειες για τη μεταφορά των δεδομένων. Για τις ρήτρες της σύμβασης υπάρχουν δύο ειδών, οι ad hoc, που είναι πολύ λίγες, και εκείνε που εγκρίνει η Κομισιόν. Οι περισσότερες μεταφορές γίνονται με βάση αυτές τις ρήτρες που εγκρίνει η Ένωση. Γι' αυτό υποχρεώνονται οι αρχές να δίνουν άδειε μεταφοράς γιατί υπάρχει απόφαση της Κομισιόν σχετική, το υπενθύμησε και ο δικαστής το δεσμευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της Κομισιόν. Αλλά οι ρήτρες αυτές προβλέπουν και τη δυνατότητα να απαγορεύσουν οι αρχές μία μεταφορά, ιδιαίτερα όταν ο νόμος, η νομοθεσία του κράτους που ενδιαφέρεται για την μεταφορά δίνει τη δυνατότητα αποκλεισμού ή εξαίρεση από τις ρήτρες αυτές πέρα των ορίων που προβλέπονται από μια δημοκρατική κοινωνία. Αν ο εισαγωγεύς δηλαδή δεν σέβεται την εθνική νομοθεσία. Άρα η Προεδρία του G29 ζήτησε από τρεις ομάδες εργασίας να συνεργαστούν για να αποτιμήσουν σε ποιο βαθμό η Αμερικανική νομοθεσία και τις πληροφορίες αυτές επιτρέπει την πρόσβαση σε δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών που προστατεύονται από την Ένωση και αν γίνονται σεβαστές οι εγγυήσει που απαιτούνται όπως τις περιγράφει ο Ευρωπαίος Δικαστής. Η ιδέα λοιπόν είναι να ορίσουμε τι θα ήταν αποδεκτή εξαίρεση σε μια δημοκρατική κοινωνία με βάση την απόφαση. Οι αναλύσεις λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα ψηφίσματά του είναι πολύ χρήσιμα ουσιώδη για μας και θα τα χρησιμοποιήσουμε. Εξάλλου η ανάλυση των δικαιοδοσιών που έχουν οι εθνικές αρχές για απαγόρευση μεταφοράς και το πώς μεταφράζονται αναέθνος γιατί δεν έχουν ακριβώς τις ίδιες δικαιοδοσίες όλα τα κράτη σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτούμε και τον τρόπο με τον οποίο θα ασκείται αυτός αυτό το δικαίωμα ελέγχου απριόρι και αποστεριόρι. Έπειτα, ο συντονισμός των προσφυγών και παραπώνων. Με ρεαλιστικό συγκεκριμένο τρόπο και τις κυρώσεις εφόσον χρειαστούν. Και βέβαια αργότερα η αποτίμηση, η αξιολόγηση της πιθανής μετατροπής αυτών των εργαλείων αν χρειαστεί να ενημερωθούν, να προσαρμοστούν γνωρίζοντας βέβαια ότι αυτό δεν είναι υποχρεωτικό ούτε θα λύσει το πρόβλημα της μαζικής επιτήρησης. Και μετά οι εξαιρέσεις. Υπάρχουν εξαιρέσεις που είναι η σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου κλπ. Αλλά πρέπει να καθοριστεί πότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι εξαιρέσεις. Η Προεδρία λοιπόν του G29 αποφάσισε να οργανώσει ακροάσεις. Στην επόμενη ολομέλειά της, την 3η 24 Νοεμβρίου, θα μιλήσει ο πρόεδρος Βάντερ Βίτ του δικαστηρίου μαζί με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών η οποία σιγά σιγά παίρνει όλη τη θέση που της αρμόζει. Η περίπτωση Σρέμς λοιπόν, η υπόθεση Σρέμς βλέπετε ότι μπόρεσε να καταλήξει σε μια δικαστική απόφαση πολύ ουσιώδη για τον πολίτη. Οι επιχειρήσεις και οι πρόσωποι τους επίσης μπορεί να συνέλθουν εκεί, γιατί πρέπει και αυτές να πάρουν μαθήματα από την απόφαση, να οργανωθούν οι επιχειρήσεις γνωρίζοντας ποιος είναι ο κίνδυνος στην περίπτωση μεταφοράς προσωπικών δεδομένων παρατύπως. Γίνεται πολλής λόγος για risk-based approach και accountability που λένε. Σήμερα αυτά θεωρούνται πολύ φλού και αγγλοσεξονικές έννοιες. Αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ χρήσιμες έννοιες. Καθώς και η αρχή της φρόνησης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνε τους λοιπόν για τη μαζική επιτήρηση και μερικές ήδη έχουν αρχίσει να το σκέφτονται. Είναι προφανές ότι η απόφαση έχει επιπτώσεις πολύ ευρύτερες από ό,τι φαινόταν στην αρχή. Μία, ένα από τα βασικά της κλειδιά είναι τι προκύπτει ως προς την μαζική επιτήρηση από τη χάρτα των θεμελιωδών. Πρέπει λοιπόν να δούμε όλες τις επιπτώσεις και προσαρμογές άλλων αποφάσεων που μπορεί να χρειαστούν όπως και σε υποθέσεις που ακόμη δεν έχουν εκδικαστεί όπως την υπόθεση Λαμπρέλα. Πρέπει να γίνει διαβούλευση με τα κράτη, με έλλη, ώστε να ληφθεί υπόψη σε όλο το νομική τάξη της Ένωσης η απόφαση αυτή. Όπως βλέπετε έχουμε κινητοποιηθεί πλήρως, γιατί παίρνουμε πολύ σοβαρά αυτή την απόφαση, ιδιαίτερα τον ρόλο μας ως εγγυητή των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων, καθώς και την ανεξαρτησία του ελέγχου των εργαλείων αυτών. Αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου και αν καταλήξουμε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα εργαλεία, τότε θα πάρουμε τα μέτρα που απαιτούνται. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας λοιπόν για τους επόμενους τρεις μήνες που θελήσαμε να σας παρουσιάσαμε, διότι η εφαρμογή αυτής της απόφασης είναι πρόκληση για όλους και η Ευρώπη δεν θα αποκτήσει αξιοπιστία στην, ως προς τις αξίες της παρά μόνον εάν αποδείξει ότι μπορεί να ελέγξει την, ιδιο, την περιπτώσει παραβίας ιδιωτικής ζωής. Μαζί σας ελπίζουμε γιατί και εσείς επενδύσατε πολύ σε αυτό ώστε από κοινού να βρούμε κλήσεις επικοδομητικές. Σας κατευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ρεϊνάλ για την έκθεση αυτή μας ε, ενημερώσατε αναλυτικά για αυτό το πολύ περίπλοκο ζήτημα. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο για τον κύριο Άλμπρεχτ που είναι και ο εισηγητής μας, αλλά δεν τον βλέπω. Εδώ ήταν, αυτή τη στιγμή όμως λείπει. Γι' αυτό θα δώσω λόγο στη σκιώδη εισηγήτρια κυρία Λορινστίν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Υποστηρίζω αυτή την απόφαση και όλη τη διαδικασία αυτή, διότι επηρεάζει πολύ τη δουλειά μας για την κανονισμό σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Σε πολλά άρθρα λοιπόν λάβαμε υπόψη την απόφαση, την διατύπωση, τις διατάξεις και κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου που λαμβάνει η χώρα θα αποτελέσει αυτό βάση για τη διασφάλιση των υψηλών στάνταρ προστασίας των δεδομένων στην Ευρώπη. Αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι αυτό το μεγάλο επίπεδο προστασίας. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ένα τέτοιο μεγάλο επίπεδο και να αντιμετωπίσουμε και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Από τη μία στιγμή στην άλλη εμφανίζονται προβλήματα πρακτικά που δεν μπορούν να επιληθούν. Το θέμα της εθνικής ασφάλειας, για παράδειγμα, είναι εκτός της δικής μας εντολής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Και βέβαια πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα τηρούνται αυτά τα υψηλά στάνταρ, διότι όλα τα όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα της έφεσης και τα λοιπά. Όμως ε, σε πολλά κρατημέλη αυτό δεν υφίσταται. Και το συζητάμε σχεδόν μετά από κάθε τριμερή διάλογο. Η ερώτησή μου λοιπόν και προς την Κομισιόν είναι πώς το λύνουμε αυτό. Πώς το λύνουμε γιατί σήμερα, μόλις σήμερα, καθόμασταν με τον εισηγητή και λέγαμε κάτι πρέπει να κάνουμε. Αν ας πούμε η κατάσταση είναι το θέμα των προσφύγων. Αν δείτε τα προβλήματα, αν δείτε πώς η μία αστυνομία από τη μία χώρα αποστέλλεται σε άλλη χώρα για να λάβει μέρος σε επιχειρήσεις, πραγματικά ε, η βάση και οι εγγυήσει, ε, ακόμα και στο δικό τους χώρο, δεν είναι ξεκάθαρα. Η απόφαση του δικαστηρίου ίσως ε, ε, να αφορά μια τρίτη χώρα, όμως δεν θα πρέπει να περιμένουμε, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να φτάσει και στα δική μας ε, πόρτα ή πρέπει να κάνουμε κάτι πριν. Ευχαριστούμε την κυρία Λοριστίν, ο κύριος Φως. Ευχαριστώ για την παρουσίαση, την οποία από τη δική μου πλευρά Μισό λεπτό να περιμένουμε τη διερμηνία. Να βάλετε τα ακουστικά. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Το δικό μου αίσθημα και από τις αναλύσεις σας ε, είναι διαφορετικό με τρομάζει λίγο ότι μέσα από μία απόφαση φτάνουμε τόσο μακριά και βγαίνουν τόσα πολλά ε, θέματα ελέγχου ε, πραγμάτων που ως τώρα δεν είχαμε καν ακούσει. Οι Γερμανοί συνάδελφοί σας, ε, οι οποίοι πήραν ένα έγγραφο με 14-20 πόσα είναι αυτά τα σημεία, πρέπει να μεταφέρουν ε, στοιχεία πάντοτε βάσει των στάνταρ και των δεσμευτικών κανόνων συνεργασίας και όλα αυτά αμφισβητούνται. Νομίζω ότι πάμε πολύ μακριά. Νομίζω ότι στην Ευρώπη δεν είμαστε ε, ε, μία νήσος ευτυχισμένων όσον αφορά τα δεδομένα. Πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών. Όσον αφορά τη μαζική ανταλλαγή, θα πρέπει να δούμε ε, ότι υπάρχει αυτή η νομική βάση, η οποία είναι επαρκής και θεωρώ ότι μάλλον πάμε πολύ μακριά και βασικά θέτουμε σε κίνδυνο όλη αυτή τη διαδικασία αν πάμε τόσο μακριά. Θα δούμε λίγο τι θα πει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, αν επικεντρωθούμε σε αυτό, ίσως ε, να μην είναι επαρκές ε, διότι δεν έγιναν οι κατάλληλοι έλεγχοι από την Επιτροπή. Η απόφαση λοιπόν αυτή για την επάρκεια είναι κάτι που θα θέσει υπό αμφισβήτηση τη βάση. Το ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις ε, της Επιτροπής για την προστασία των δεδομένων. Αυτό έπρεπε να έχει ελεγχθεί αλλά και τα εργαλεία που ε, υπάρχουν στην οδηγία και σε αυτό δεν πρέπει να τίθενται σε αμφισβήτηση και αναρωτιέμαι γιατί εσείς το κάνετε αυτό. Και οι συνάδελφοι από τη Γερμανία αντίστοιχα. Δηλαδή στην ουσία ε, απομακρυνόμαστε από τη μαζική μεταφορά δεδομένων και αυτό δεν είναι πραγματικά κάτι που συνάδει με το πνεύμα που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Σε επίπεδο βάσης ε, νομικής ίσως να είναι πολύ σημαντικό αυτό το ε, βούλευμα. Ο, ας πούμε για τους γάμους, αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό, αλλά το να πετάμε, να μαζί με τα χλωρά να καίγονται και τα ξερά, ε, τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά δεν είναι σωστό. Και Τώρα λέει πρώτος να δώσουμε το λόγο στην τελευταία σκιωδησγήτρια είναι η κυρία Έρστ. Έχετε το λόγο. Νόμιζα ότι πάμε αναομάδα, αλλά δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ. Θα ρωτήσω άλλη μία φορά. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το θεωρώ ότι είναι σημαντικό να το πούμε με για το γεγονός ότι έχουμε πολύ συγκεκριμένη εικόνα και έχουμε ακούσει τόσο συγκεκριμένα πώς έγιναν όλα αυτά. Ήθελα απλώς να ξεκαθαρίσω το εξή μετά την απόφαση τώρα, τι χρειαζόμαστε στην πραγματικότητα, χρειαζόμαστε μια καλύτερη διαδικασία, μπορούμε με τους binding corporate rules και τα standard contract ε, clauses να ξεκινήσουμε να βρίσκουμε κάτι που είναι λύση. Μπορείτε λίγο να μας το ξεκαθαρίσετε αυτό. Και σε τι βαθμό χρειάζεται ό,τι χρειάζεται. Υπάρχει αυτή η παραδοσιακή ιστορία με τη μαζική παρακολούθηση που γίνεται συνεχώς και τρέχει και τρέχει και νομίζουμε ότι είμαστε και το ε, πιο ασφαλές μέρος που ελέγχεται πάρα πολύ καλά, όμως ε, τελικά τα δεδομένα και τα στοιχεία της αστικής ασφάλειας συγκεκριμένων αρχών τελικά με... βγαίνουν παρά έξω. Τέλος. Μιλήσατε για το PNR, το TTIP. Μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα γι' αυτό. Ε, υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να υπάρχουν στην ακρόαση. Και επίσης υπάρχει και η επιρροή αυτής της απόφασης σε άλλους ευρωπαϊκούς νόμους και συμφωνίες κτλ. Μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Τσίπελ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την έκθεση. Από τη στιγμή που ελέγχουμε κατά πόσο γίνεται μια σωστή ε, μεταφορά δεδομένων, μπορούμε να μεταφέρουμε τα δεδομένα, αλλιώς όχι. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε σε τι επίπεδο υπάρχει προστασία δεδομένων και όσον αφορά και στους ελέγχους ε, παραμένει σημαντικό να υπάρχουν αυτά τα δύο επίπεδα. Πρώτον, η κανονική νομοθετική διαδικασία και να τηρούνται συγκεκριμένα στάνταρα από τις επιχειρήσεις και το άλλο είναι το θέμα των μυστικών υπηρεσιών τι ε, δεδομένα έχουν αυτές και νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα ευρωπαϊκό στοιχείο. Τα, οι μυστικές μας υπηρεσίες ε, πάντοτε έχουν πρόβλημα αν εμείς ελέγχουμε τι ακριβώς έχουν ως αρμοδιότητα και τι άδεια έχουν. Για, ε, για διάφορες συμφωνίες όπως την TFTP και τα λοιπά θα ήταν καλό ε, τουλάχιστον έμεσα ε, να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, ας πούμε για μια ευρωπαϊκή συμφωνία για τα δεδομένα των επιβατών σε πτήσεις να δούμε τι γίνεται και με τις τρίτες χώρες αν τέλος πάντων θίγονται και αυτές και φυσικά υπάρχει και το θέμα της εθνικής ασφάλειας όταν υπάρχει ένα εθνικό ζήτημα θα πρέπει να το αξιολογούμε πολύ προσεκτικά, να υπάρχουν συγκεκριμένες νομοδοτήσεις ε, και να γίνεται εντατική εργασία από τις υπηρεσίες ε, και από ε, διεθνείς φορείς που ασχολούνται με την ασφάλεια. Το γεγονός λοιπόν ότι πρέπει να δούμε κατά πόσο επηρεάζονται και οι ευρωπαϊκές ε, συμφωνίες είναι κάτι που πρέπει να ελεγχθεί. Ευχαριστούμε την κυρία Τσίπελ. Ο κύριος Κύρκο έχει το λόγο. Είστε και εσείς ε, εισηγητής ε, σκιώδης από την ομάδα ECR. Σε ευχαριστώ και συμπαθάτε με που έλειψα για λίγο και δεν άκουσα το πρώτο τμήμα γιατί διάβασα με ενδιαφέρον το έγγραφο της ομάδας εργασίας και ήμουνα στις ε, είπα στην ακρόαση του Κογκρέσου για τα θέματα του Safe Harbor και αυτό σχετίζει με τα συμπεράσματα στα οποία ε, συμπυκνώθηκε η υπόθεση Σρέμς. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε να καταλήξετε σε κάποιο είδους ε, ρήτρες διαφύλαξης, σε κάποιο είδους ε, συμπεράσματα για τα δεδομένα που αυτό θα είναι πολύ χρήσιμα ε, ε, από εμπορική πλευρά για τι σχέσει ε, ΕΠΑ Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ερωτώ τα εξή. Όσον αφορά το θέμα τη απόφαση και εάν θεωρήσουμε ότι θα υπάρξει ικανοποιητική κατάληξη, θεωρείτε ότι θα έχει ένα δρομικό χαρακτήρα αυτή η απόφαση και σε ποιο βαθμό Επίσης σε ποιο βαθμό θα επιδέχεται ένδικα μέσα αυτή η απόφαση. Θα έχει εκτελεστό χαρακτήρα. Ή τα γεγονότα το έχουν ξεπεράσει ήδη. Και υπάρχει κάποια διαδικασία ε, στο ΔΕΚ που να επιτρέπει κάποιο είδους ε, έφεση ή κάτι συναφές. Κάτι άλλο τώρα. Ενώ έχουμε, είπαμε, στην εργασίας. εναλλακτικέ ε, αν δεν υπάρξει το safe harbor. Μπορεί να εξετάσει η εργασία τα διαφορετικά αποτελέσματα για τους διαφορετικούς κλάδους εμπορικής και επιστημονικής δραστηριότητας. που εγώ κατάλαβα. Υπάρχουν μέσα εναλλακτικά τα οποία αφορούν μεγάλες εταιρείες. Εκείνες που έχουν την οικονομική δυνατότητα να φέρουν το οικονομικό βάρος αυτών των ε, μέσων. Εάν τα πράγματα εξελιχθούν όπως προτείνεται και υπάρξει τελικά κάποια συμφωνία, τι άλλο θα μπορούσε να απασχολήσει σαν θέμα προτεραιότητας την ομάδα εργασίας. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο, Πρόεδρος. Ο επόμενος. Ευχαριστώ. Εκτιμώ ιδιαίτερα την παρουσίαση που έγινε και την ανάλυση των επιπτώσεων αυτής της σημαντικότατης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εσείς ήρθατε για να μιλήσετε για το εβδομάδα εργασίας του άρθρου 29. Το άρθρο αυτό δείχνει ότι η οδηγία για την προστασία των δεδομένων ζει ακόμα. Και λυπάμαι γι' αυτό γιατί θα ήθελα αντί για αυτή την οδηγία να υπήρχε ήδη Data Protection pack Το νέο, η νέα δέσμη προστασίας δεδομένων που επίκειται αλλά εφόσον δεν έχουμε ακόμα αυτό το νομοθέτημα που επεξεργαζόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια, ισχύει ακόμα η οδηγία για την προστασία των δεδομένων και εσείς εκπροσωπείτε μια ομάδα εργασίας που αποτελείται από εκπροσώπους όλων των μελών της Ένωσης που ασχολούνται με την καθημερινή εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Αυτό ήθελα να προσθέσω στη συζήτησή μας. Φυσικά συμβαρίζομαι τις περισσότερες ανησυχίες που ακούστηκαν. Η δική μου όμως είναι αφορά το αποτέλεσμα που θα έχουν όλα αυτά πάνω στη ζωή των χωρών μελών, διότι η απόφαση αυτή δεν αφορά μόνο τις διμερείς σχέσεις Ένωσης με Ηνωμένε Πολιτείες μέσω της λεγόμενης ε, συμφωνίας του ασφαλούς λιμένα που ακύρωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επίσης επηρεάζει και όλες τις άλλες διμερείς συμφωνίες της Ένωσης με τρίτες χώρες εφόσον υπάρξει αυτή η δεσμευτική ερμηνεία του δικαστηρίου για τη χάρτα των θεμελιωδών. και θα έχει την ίδια ισχύ περίπου με το πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης αλλά επίσης επηρεάζει και τα νομικά συστήματα όλων των χωρών μελών τα εθνικά που κυρίως εκπροσωπεί η ομάδα εργασίας του άρθρου 29. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν πώς αναλύεται την επίπτωσή της στα εσωτερικά εθνικά νομικά συστήματα για τις μεταφορές δεδομένων που γίνονται από τις χώρες μέλη σύμφωνα με λανθασμένα πρότυπα. Πώς θα αναθεωρηθούν με υπό το νέο φως αυτής της απόφασης του δικαστηρίου που είναι πιο απαιτητική από ποτέ. Δεύτερον, τι προβλέπετε ως επίπτωση όχι μόνο για τις μεταφορές δεδομένων αλλά και για τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που, που, που, που, που, που λέω θα ελέγχονται στο εξής περισσότερο με βάση την χάρτα των θεμελιωδών και ρήτων, Η μαζική επιτήρηση που κάνουν κράτη-μέλη. Τι θα γίνει. Υπάρχουν τέτοιες επιτηρήσεις από τα κράτη-μέλη και ποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μήπως μερικές χώρες μέλη ιδιαίτερα, ιδιαίτερα θα ελεγχθούν για κάποιον ειδικότερο λόγο από ό,τι ξέρετε, από ό,τι είδατε υπάρχει κανένα κράτος που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Με βάση λέω τη χάρτα των θεμελιωδών λέω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Λόπες Αγγιλάρη, πριν δώσουμε το λόγο στην εισήτρια μας, παρακαλώ, εάν θέλουν τους εκπροσώπους Κομισιών και Συμβουλίου να λάβουν το λόγο. Υπάρχει κάποιος. Κομισιόν, Συμβούλιο. Καλά. Σας δίνω το λόγο κύριε. Πρώτα πρώτα σας ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις. Έτσι αποδεικνύεται ότι πραγματικά ενδιαφέρεστε και ότι χρειάζεται να γίνουν κάποιες μεταβολές αναγκαίες για αυτό το θέμα το οποίο είναι τόσο λεπτό και δύσκολο και στους 29 αλλά και ότι θα πρέπει κανείς να συζητήσει και ενδεχομένως να αλλάξει απόψεις. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ για τις τόσο ενδιαφέρουσες και εύστοχες ερωτήσεις. Επίσης, για να τα πάρουμε με τη σειρά. Υποβολή των ερωτήσεων. Πρώτα-πρώτα. Η προβληματική της εθνικής ασφαλείας. ότι πολλές φορές αυτά τα θέματα είναι εκτός αρμοδιότητας των θεσμών. Όντως. Και στο G29 έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την δυσκολία όσον αφορά την ανταλλαγή των ομολόγων, γιατί πολλέ φορέ και εμένα και δεν είμαι θα αρμόδιο σε επίπεδο υπηρεσιών ε, πληροφοριών. Οπότε υπάρχουν κάποιες αρχές που έχουν βρει ε, ε, πεδίο αρμοδίζων, άλλες όμως όχι. Και αυτό πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις από αυτών των θεμάτων που είναι τόσο λεπτάκι δύσκολο για να σας δώσω δε ένα παράδειγμα Έχουμε το νόμο 318 που μεταφέρει την οδηγία του 95, ο οποίος αφορά τις υπηρεσίες ασφαλείας. Κατόπιν δε έχουμε διάφορες ε, ρυθμίσεις, αλλά η υπηρεσία πληροφοριών είναι αρμόδια επί τη βάση κάποιων κανόνων που έχουν κάνει τις πληροφορίες, αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Οπότε δεν ενημερώνονται για την ύπαρξη κάποιων θεμάτων, κάποιων φακέλων. Η ΚΝΙΝ αυτά. Οπότε είναι δυνατόν να υποβληθεί έτοιμο από το, από το Γαλλικό Κοινοβούλιο. Αλλά αυτό δεν μπορεί να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Ε, Επίση, από πλευρά των εκτοστέρων ελέγχων, η ΚΝΙΛ μπορεί να ασκήσει έλεγχο, αλλά όχι για όλα τα θέματα. Μπορεί να επιβάλλει γύρω αλλά όχι για όλα. Οπότε υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις που έχουμε επιφέρει για αυτά τα θέματα πληροφοριών και επίσης ε, ε, όλα αυτά είναι χρήσιμα και για άλλες ε, αρχές. Στο g συμμετέχει η πρόεδρος του ΚΝΙΛ και πολλές φορές ζητεί σε εθνικό επίπεδο περισσότερες αρμοδιότητες ελέγχου των και εκ των υστέρων για αυτά τα θέματα και με την ευκαιρία να σας πω ότι στη Γαλλία έχουμε κάτι που λέγεται δικαίωμα άμεση πρόσβαση. Αυτό το σύστημα λειτουργεί καλά για ε, όλα τα, τα δημόσια θέματα και φάκελους ούτως ώστε μπορούμε αυτό το σύστημα να θέσουμε κάτι στην κνήλη η οποία θα πάει και θα επαληθεύσει και θα διαπιστώσει κατά πόσο η επεξεργασία ε, των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον νόμο. Δεν λέμε ότι πρόκειται να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος, βέβαια. Αυτό θα ήταν αντιφατικό, αλλά μπορεί να ε, ελέγξει, να διασταυρώσει, να δει κατά πόσο είναι σύνομα όλα αυτά και να το επισημάνει. Ίσως να επιβλαβάλλει κάποιο καιρό. Λοιπόν, βλέπουμε και κάτι σαν αντίβαρο που υπάρχει και επίσης με αυτό το ζήτημα του ελέγχου από το ε, Συμβούλιο Επικρατείας και το Συνταγματικό Δικαστήριο. Οπότε έχουμε κάποια συστήματα σε εθνικό επίπεδο και αλλού εκτό από τη Γαλλία. Αλλά είναι περίπλοκο το πώ τελικά θα υπάρξει εναρμόνιση αυτών των πρακτικών και του ελέγχου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Επ' αυτού θα ασχοληθεί το G29 για τα διάφορα εθνικά συστήματα τόσο ώστε να υπάρχει σύγκριση και να δούμε πώς θα υπάρχει ο έλεγχος και θα δούμε τι μέσα προσφυγής ε, έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες για το δεύτερο ερώτημα τώρα. Ότι έχουμε ευρεία ερμηνεία της απόφασης και για τα άλλα εργαλεία μεταφοράς και διαβίβασης των δεδομένων στην Ευρώπη. επισημαίνουμε δύο τινά. Σήμερα δεν λέμε ότι αυτά τα εργαλεία πλέον δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή ότι δεν συνάδουν προς ό,τι απαιτείται για την Ευρώπη. Όμως θα κάνουμε κάποια ανάλυση αυτών των εργαλείων και θα δούμε κατά πόσον, ε, σύμφωνα με την απόφαση, υπάρχουν οι κατάλληλες εγγύσεις για τη χρήση αυτών των εργαλείων. Γιατί Πρώτα πρώτα, νομική απάντηση, διότι στις ε, ε συμβατικές ρήτρες έχουμε το άρθρο 4, για κοιτάξτε, και εκεί τίθεται κάποια προπόση, ότι δηλαδή οι αρχές απαγορεύουν τη διαβίβαση των δεδομένων, άπαξ και υπάρχει ένας αλλοδαπός νόμος ο οποίος ορίζει αυτός ο οποίος θέλει τα δεδομένα να μπορεί να παρεκκλίνει από το κοινωτικό δίκαιο. Άπαξ και αυτή η παρέκκληση αντιβαίνει προς όσα ισχύουν στο κράτος εκείνο. Επομένως, χρησιμοποιούμε τα κριτήρια της απόφασης. Και άρα, φυσιολογικά το ερώτημα, εάν για την απόφαση θα πρέπει να κρίνει ο δικαστής, ε, εάν είναι αποδεκτό να υπάρχει κάποια παρέκκληση. Και αυτά είναι τα κριτήρια, δηλαδή το κατά πόσον τα εργαλεία αυτά περιβάλλονται από τις δέουσες εγγύησεις. Από τη θυμάμαι, ε, περί, περί την παράγραφο 90 της απόφασης τοποθετείται ο δικαστής για το επίπεδο της ε, προστασίας, για το, το κατά πόσο είναι αρκετό το επίπεδο προστασίας της ΣΥΠΑ και επομένως θα πρέπει και οφείλει να το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άπαξ και υπάρχει τέτοιου είδου διαπίστωση. Να κάτσει δηλαδή και να δει τι ισχύει και στην Αμερικανική Ένωμη Τάξη και κατά πόσον ε, θα τηρεί το κοινοτικό δίκαιο όποτε έχουμε το δεδομένα προς τους Αμερικανούς. Οπότε είπαμε θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Το θέμα δεν είναι να μπλοκάρουμε πάσα διαβίβαση δεδομένων προς τις ΗΠΑ, ΕΕ, διότι γνωρίζουμε για τις επιπτώσεις που θα είχε κάτι τέτοιο από πλευράς οικονομικής. Γι' αυτό και έχουμε φτιάξει αυτή την φούσκα ε, της μεταβατικής περίοδου του τριμήνου. Οπότε επιτρέψαμε στα κρατημένα να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία. Οπότε και λάβαμε κάποιους κινδύνους σχετικά με αυτή την κίνηση. Όμως είπαμε θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Και επίσης καθόμαστε και ζυγίζουμε τις συνέπειες. Η απάντηση θα δοθεί εδώ και τώρα, αφού στα σοβαρά, ενδελεχώς, κάτσουμε και σκεφτούμε ποιο είναι το νομικό πλαίσιο, ποιες είναι οι παρεκκλήσεις, θα δούμε τι γίνεται με το άρθρο 4, εάν δεν πληρούνται οι όροι του ή ου. Αυτό ήταν το δεύτερο θέμα. Το τρίτο τώρα. Τι χρειάζεται. Είναι το ερώτημα το οποίο ανακύπτει γιατί όπως έλεγα για το πρωτοτοπίο στο G29. Κάθε φορά που συζητούμε την υπόθεση αυτή, η απάντηση δεν είναι στα συμβατικά εργαλεία. Δεν είναι στο πόσο θα τα αναβαθμίσουμε. Άπαξ και αυτά τα εργαλεία δεν επηρεάζουν το νομικό πλαίσιο για κάποιον που θα αναδεχθεί τις πληροφορίες. Εάν λένε τα εργαλεία αυτά ότι θα πρέπει να τηρήσουμε τα στάνταρ και τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αν επιβάλλεται η τήρηση των όσων λέγονται εκεί για αυτόν που θα λάβει τις πληροφορίες άπαξ και το νομικό πλαίσιο του εισάγοντος τις πληροφορίες ε, δεν το επιτρέπει ναι. συμμορφωθεί προς το κοινοτικό δίκαιο αλλά και το σύνολο των ε, συμβατικών ρητρών τότε υπάρχει πρόβλημα πρόβλημα ιεραρχίας κανόνων δικαίου επομένως για αυτό το λόγο θα πρέπει να χωνέψουμε τι ισχύει και να αναγνωρίσουμε ότι η λύση έγκυται αλλού και θα προέλθει από μια διακυβερνητική συμφωνία λαμβάνοντας υπόψη τις ε, ευρωπαϊκές αρμοδιότητες, κομισιόν, κράτη-μέλη, μια συμφωνία που θα έχει επαρκή νομική ισχύ και έτσι να μπορεί ο εισάγων τα, τις να συμμορφώνεται με το κοινωτικό δίκαιο. Άρα η λύση δεν είναι ούτε εύκολη ούτε αυτονόητη. Παρακάτω. Όλοι εμπλεκόμενοι να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται και όλων γίνεται περισσότερη κουβέντα για αυτά. Επιχειρήσεις, κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει να υπάρξει τελικά συμφωνία που να οργανώνει τη συνεργασία ε, επί των πληροφοριών αυτών. Ποιος κάνει να υπάρξει τελικά μια ρύθμιση που να καλύπτει όλα τα θέματα. Όχι να πούμε ότι δεν υπάρχει πλέον πρόσβαση, δεν επιτρέπεται ούτε μία παρέκκληση. Ναι, επιτρέπεται η παρέκκληση, αλλά αυτή η παρέκκληση θα πρέπει να ρυθμιστεί με κάποια κριτήρια. Δικαστικά, ενδικά μέσα, διαφάνεια, αναλογικότητα, ε, σκοπιμότητα, του τι χρειάζεται δηλαδή. Αυτά θα πρέπει να λαμβάνει ο δικαστής υπόψη. Αυτά για το τρίτο ερώτημα. Τέταρτο. Για όλα αυτά που έχουν σχέση με το TTIP και τις άλλες διατλαντικές συμφωνίες. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για τις άλλες δηλαδή διεθνείς συμφωνίες. Και εδώ θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες για τα άλλα εργαλεία. Δηλαδή, να μην μόνο δεν υπάρχουν συνέπειες, αλλά να κάτσουμε να προβληματιστούμε για αυτές τις συνέπειες. Τι να σας πω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Οι ελεκτικές αρχές του G29 θα πρέπει επίσης να προβληματιστούν για τις ενδεχόμενες συνέπειες αυτές. Τώρα, όσον αφορά τις εναλλακτικές, και τα αποτελέσματα για τις διάφορες επιχειρήσεις, για τις νέες συμφωνίες, για αν υπάρξουν. Εν μέρει απάντησα. Κυρίως για το θέμα των εγγύσεων που θα πρέπει να παράσει μια τέτοια συμφωνία. Δυνατότητα ενδίκων μέσων, διοικητικών κλπ. Τι είναι σκόπιμο να υπάρχει διαφάνεια. Όλα αυτά θα πρέπει να πλησιώνονται από τις εγγύσεις για την ε, διαβίβαση και χρήση των ε, πληροφοριών. Το θέμα δεν είναι το τι θα μπει σε αυτή τη συμφωνία, γιατί έχουμε την απόφαση, έχουμε και ένα σωρό νομολογία του ΔΕΚ και της Επιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά θα πρέπει κάθε παρέκκληση να είναι αποδεκτή από ένα δημοκρατικό καθεστώ. δημοκρατική ένωμη τάξη. Άρα δεν είναι το τι θέλουμε να καλύπτει η συμφωνία, είναι το τι μορφή θα πρέπει να έχει αυτή η συμφωνία, ούτω ώστε να λειτουργεί. Να, ποιο είναι το αληθε. ερώτημα που τίθεται. Παρακαλώ. επίπτωση στα, σε άλλες νομιστάξεις και αυτό νομίζω επίσης εν μέρη το εκάλυψα. Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί βρισκόμαστε μόλι στην αρχή αυτή τη διαδρομή. Τώρα ξεκινήσαμε αυτή τη διαδρομή. Και όπω σα είπα, είναι τεράστιο ο. Τεράστιος, τα, τα περιθώρια στα οποία πρέπει να κινηθούμε. Ε, να δούμε τι θα Έχουμε τώρα τις ρήτρε, είναι για μα είναι βέβαια κάτι το κατεπήγον. Στη συνέχεια θα δούμε ποιε θα είναι οι συνέπειε τη απόφαση για άλλες αποφάσεις, για άλλα συστήματα. <coughs> Αλλά για μια φορά δεν μπορούμε τώρα να εξαγάγουμε όλα τα συμπεράσματα και θεωρούμε ότι σε σχέση με το βεληνικές αυτής της απόφασης δεν πρέπει να στροφοκαμιλίζουμε, να βάζουμε στην άμμο το <coughs> κεφάλι και να πούμε ότι βρέξει σας κατεβάς. Άρα θα πρέπει να δούμε το πώς θα πλαισιώσουμε αυτή τη διαβίβαση δεδομένων στο εξωτερικό. Και εάν επαρκούν τα εργαλεία θα δούμε, θα κάνουμε υπό το φως της απόφασης. Ευχαριστούμε για όλες τις επεξηγήσεις και για τα δεδομένα που μας δώσατε. Η γραμματεία μας λέει ότι οι εκπρόσωποι της ομάδας 29 θα μας επισκεφτούν άλλη μια φορά τέλη Ιανουαρίου για να δούμε τα αποτελέσματα και τις απαντήσεις στα ερωτήματα που προέκυψαν και που θα προκύψουν όπως εξελίσσεται το ζήτημα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, το σημείο 24. Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκών τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, σπουδές, συνταλλαγή μαθημάτων. Είναι το μόνο, ε, το μόνο έγγραφο το οποίο ακόμα είναι υπό διαπραγμάτευση σε επίπεδο μετανάστευσης, άτυπης μετανάστευσης. Η κυρία Σεσίλια Βίκστροπ είναι η εισηγήτρια και θα μας εξηγήσει σε ποια φάση είναι διαπραγματεύσεις. Έχετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, φαίνεται σαν να φεύγουν όλοι από την αίθουσα, αλλά με χαρά μου θα σας αναγγείλω ότι υπάρχει αυτή η έκθεση που μπόρεσε να συνταχθεί μετά από ώρες ατελείωτες διακαπραγματεύσεων και τώρα έχουμε μια πολιτική συμφωνία, ένα πακέτο για την οδηγία, για τους ε, φοιτητές, ε, τους μαθητές ε, και τους ερευνητές. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε την Τρίτη, στον τριμερή διάλογο, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, να έχουμε μια τελική έκδοση του κειμένου, για το οποίο ήδη υπάρχει πολιτική συμφωνία. Με αυτή την ευκαιρία λοιπόν να ευχαριστήσω όλους όσοι έχουν εμπλακεί σε αυτό το έργο. Εδώ και τρία χρόνια σχεδόν μεγάλο και δύσκολο το έργο και φοβόμουν ότι θα κολλήσει και για τα επόμενα χρόνια, για πολλά χρόνια στο Συμβούλιο. Μάλιστα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σχεώδεις και το προσωπικό τους γιατί πραγματικά ήμασταν εξ αρχής μια εξαιρετική ομάδα και μέχρι το τέλος παλεύαμε μαζί για τους ίδιους στόχους. Να ευχαριστήσω επίσης και το εξαιρετικό προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ τους λόγους Ρόσφρα και Ντανιέλ την βοηθό μου και στις δυο σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και για την αφοσίωσή σας σε, όλη, σε όλη τη διαδικασία. Να ευχαριστήσω επίσης την Κομισιόν για τις άοκνες προσπάθειες να μας εξηγήσουν και να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις και το Συμβούλιο για την καλή συνεργασία τους σε μια σειρά προεδριών, εκ των οποίων η Προεδρία του Λουξεμβούργου πραγματικά έδειξε μεγάλη φιλοδοξία, δημιουργικότητα και εξαιρετική συνεργασία. Είχαμε πολλές δύσκολες συζητήσεις, αλλά η συνεργασία ήταν πάντοτε εξαιρετικά επικοδομητική να εξηγήσω τις γενικές γραμμές του πακέτου. Καταρχάς είναι ένα πακέτο με μεγάλη προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη. Θα αυξηθεί το πεδίο, θα επεκταθεί για να περιλάβει τους ε, φοιτητές, τους ερευνητές, τους εκπαιδευόμενους και τους εθελοντές στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, Εθελοντικής Εργασίας. Ε, θα αυξηθεί η κινητικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ανθρώπους αυτούς και τις οικογένειές τους τα μέλη της οικογένειάς τους θα έχουν το δικαίωμα εργασίας όσο βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι φοιτητέ θα έχουν και αυξημένη πρόσβαση στην αγορά εργασία. Επίση, τώρα εισάγουμε ένα σύστημα που επιτρέπει στου φοιτητέ και του ερευνητέ να μείνουν στην Ευρώπη τουλάχιστον 9 μήνες νόμιμα εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις μελέτες και τα ερευνητικά τους ε, έργα είτε για να βρουν δουλειά, είτε για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν πλήρως την εκπαίδευση που τους παρήχαμε και για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτά τα δημιουργικά και τα λαντούχα μυαλά στην Ευρώπη, για να βοηθήσουμε την οικονομία μας. Οι ΟΠΕΡ επίση, οι εσωτερικές δηλαδή, θα μπορούν να υποφεληθούν κατ' επιλογή. Είναι η πρώτη φορά που περιλαμβάνονται σε ένα νομικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε γενικές γραμμές λοιπόν η νέα οδηγία θα βοηθήσει τους ταλαντούχους να έρθουν στην Ευρώπη και να χτίσουν μαζί μας ένα πιο ισχυρό μέλλον, να προωθήσουν την ανάπτυξη και την ευημερία για όλους. Για να διασφαλιστούν όλα αυτά τα θετικά, επίσης φυσικά συμφωνήσαμε και σε μια σειρά δικλείδων ασφαλείας που ε, θα διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει κατάχρηση όπως λένε τα κράτη-μέλη. Κατάλληλα μέτρα για την ε, πρόληψη των καταχρήσεων. Γνωρίζουμε τα γραφειοκρατικά βάρη που υπάρχουν στα κράτη-μέλη τα οποία τα θέλουν πολύ τα κράτη-μέλη, όμως τελικά καταφέραμε να έχουμε ένα καλό συμβιβασμό. Υπάρχουν κάποια σημεία που μας αρέσουν και άλλα που μας αρέσουν λιγότερο. Τα θετικά όμως υπερτερούν σε σχέση με τα αρνητικά. Σε αυτή την ε, φάση όλοι μας έχουμε επικεντρώσει τις προσπάθειες στην επίλυση της εξίας δύσκολης κατάστασης που υπάρχει για τους ε, πρόσφυγες που φτάνουν στις ακτές μας. Τα θεσμικά όργανα λοιπόν ε, με αυτή την οδηγία θα μπορέσουν να προωθήσουν και ε, φιλόδοξες προτάσεις νομοθετικές στο θέμα της άτυπης μετανάστευσης. Κάτι που στη Βαλέτα αύριο στην Σύνοδο Κορυφής θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα νομίζω. Να ευχαριστήσω όλους όσοι, όσοι συμμετείχαν σε αυτή την έκθεση Χρειάζεται βέβαια να γίνει κάτι ακόμα για να ολοκληρωθεί το κείμενο μέχρι την Τρίτη, αλλά τότε θα τελειώσει και πιστέψτε με θα γιορτάσουμε κιόλα. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε για την υπομονή και το ενδιαφέρον που δείξατε για αυτή την έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Βίκστρομ, δυστυχώς η Σκιώδης δεν είναι εδώ. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τη γνώμη τους. Κάποιος άλλος όμως που θα ήθελε να μιλήσει. Όχι. Να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα, το 25. Η κυρία Τσινίτση είναι η συγγήτρια στην πρόταση οδηγίας για τις διασυνοριακές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτα ή κατηγορούμενα στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Είμαστε στη φάση διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο βάσει του τριμερούς διαλόγου που έγινε στις 27 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ Πρόεδρε για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για αυτόν τον τριμερή διάλογο τελευταίος που έγινε όσον αφορά τις δικονομικές εγγυήσεις για ύποπτους και κατηγορούμενους ανηλίκους. Το εσπέρο, το εύχομαι μόλι μου την ψυχή μια που δουλέψαμε τόσο εντοπικά και ελπίζω έτσι να ε, συναθεί τελικά κάποια συμφωνία. Βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη φάση πάντως τώρα γιατί στην αρχή του τριμερούς διαλόγου προέβημεν σε κάποια επιλογή δηλαδή πρώτα που θα συζητήσουμε με τα άρθρα εις τα οποία θεωρήσαμε ότι ε, δεν θα υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Πρώτα εκεί και κατόπιν να προχωρήσουμε και να στέσουμε προσοχή μας στα, άρθρα εκείνα τα οποία απαιτούν ε, μια αντιπαράθεση πιο σοβαρή, ε, μια διαφωνία πιο μεγάλη για να δούμε πώς μπορούμε να άρουμε δυσκολίες και εμπόδια γενικώ, επομένως για άλλη μια φορά βγήκανε πάρα πολλά εμπόδια και στην τελευταία τριμερή συνάντηση Γι' αυτό γιατί από πλευρά κάποιων κρατών μελών υπήρξε πάρα πολύ κλειστή αμυντική στάση και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες της Λουξεμβουργενής Προεδρίας που πάσχεσε πάρα πολύ ούτως ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες πριν το τέλος του έτους. Οπότε και εγώ και το επιτολείο μου ε, προς τα εκείνη κατεύθυνση δουλεύουμε και ευχαριστώ και τους ε, σκιώδεις εισηγητάς εδώ βρισκόμαστε τώρα, εν ώψη τη 12η του μηνό, την 5η που θα γίνει η επόμενη συνάντηση. Ευχαριστώ και τη γραμματεία μα που μα βοηθά σε αυτό το έργο που είναι τόσο δύσκολο σε αυτή την τελευταία φάση. Αλλά θα πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει όμως να είμαστε ικανοποιημένοι για όσο πετύχαμε μέχρι τώρα. Κλείσαμε τη συμφωνία για πολλά άρθρα. Να, να σας αναφέρω μερικά από αυτά τα πιο σημαντικά. Φερρυπίν. 15. Εκεί πετύχαμε να εντάξουμε το δικαίωμα του ανηλίκου να συνοδεύεται από τον έχοντα την ε, επιμέλεια ή σε όποιον ανατεθεί αυτό. Και όχι μόνο ε, όταν ε, παρίσταται στο ακροατήριο, αλλά και σε άλλες φάσεις. Οπότε αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και διότι είχαμε να κάμψουμε την στεναρή αντίσταση του Συμβουλίου. Αλλά και γιατί δεν προβλεπόταν μια τέτοια ρύθμιση ούτε στην προσέγγιση που γινόταν ούτε στην αρχική στάση του Συμβουλίου. Άρα καλά τα πήγαμε σε αυτό το σημείο. Το ίδιο ισχύει και για ένα άλλο σημείο. Άρθρο 8. Δικαίωμα σε ιατρική εξέταση. Και εδώ καλύψαμε και το δικαίωμα εις ιατρική αρρωγή. Ευρύτερο αυτό του πρώτου. Ούτε αυτό προβλέπονταν στην αρχή πρόταση της Κομισιόν. Οπότε γι' αυτό σας λέω ότι και αυτό είναι σημαντικό και αποδεικνύει πόσο καλά τα πήγε το Κοινοβούλιο. Πόσο καλά τα πήγαμε στην τριμερή αλλά έχουμε και κάποια άλλα θέματα τα οποία συζητούνται και πάνω σε αυτά θα πρέπει κάπου να καταλήξουμε 10, 11, 12 τα άρθρα αυτά να παραταθούν όλες οι εγγύσεις σε όλους τους α, ανηλίκους που τους στερείται η ελευθερία. Όχι μόνο σε εκείνους που είναι σε φυλακή. Θα πρέπει σε αυτό κάπου να καταλήξουμε βεβαίω και υπάρχει δυσκολία, αλλά επί των εγγύσεων. Υπάρχει καταρχήν συμφωνία όμως καταβάλλεται κάποια προσπάθεια να υπάρξει παρέκταση αυτών των εγγύσεων. Όχι μόνο για τους κυριολεκτικά κρατουμένους. Είχαμε μια τεχνική συνάντηση και θα δούμε αν στην επόμενη τριμερή συνάντηση θα τα βρούμε. Ελπίζουμε ότι η ιδιωτικότητα του βίου των ανηλίκων θα αναγνωριστεί επίσης και οι εγγυήσεις σε σχέση με την ανάκριση των ανηλίκων. Πάντως, ακόμα το δύσκολο σημείο είναι το άρθρο υπαριθμών 6 για το δικαίωμα εις την υπεράσπιση. Και να δούμε τι θα γίνει με το πεδίο εφαρμογή οδηγία σχέση με αυτό. Μιλούμε για ανηλίκους. Έχω προσωπική εμπειρία, έχω δουλέψει αυτά τα θέματα. Μιλούμε για ανηλίκους και πολλές φορές θεωρούμε τα πράγματα είναι πιο εύκολα και δεν είναι όμως στην πραγματικότητα για εξού και οι δυσκολίες αυτές και γι' αυτό και θέλουν να υπάρχουν αυτές οι εγγύσεις ενσωματωμένες στο κείμενο είναι σημαντικά αυτά και βέβαια όλα αυτά ισχύουν και κατά αναλογία και ή θα μπορούσαν να ισχύουν και για τους ενηλίκους Είπαμε επομένω ότι πού είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα και άρα, συνοψίζοντας, τα βασικά προβλήματα είναι από την αμυντική του Συμβουλίου σε σχέση με το τι θέλουν να προβλέψουν για του ανηλίκου όσον αφορά την υποχρεωτική παρουσία του συνηγόρου. Επίση, το ότι θα θέλουμε να υπάρξει κάποιο είδου ε, σύνδεση με την οδηγία που προβλέπει την πρόσβαση σε δικηγόρο. Το πρόβλημα είναι ότι η οδηγία αυτή περιέχει μία σειρά από παρεκκλήσεις που οπωσδήποτε δεν είναι παραδεικτές. Δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει αποδεκτό σε κάποια οδηγία για τους ανηλίκους. Οπότε όλα αυτά μας οδηγούν στο να σκεφτούμε ότι χρειάζεται η αυξημένη προστασία των ευαλώτων ανηλίκων. Μιλούμε για υπόπτους και μιλούμε και για κατηγορουμένους, αλλά η απενική διαδικασία και αυτό και πρέπει να είναι πιο ψηλή, πιο μεγάλη προστασία. Άρα θα πρέπει να δούμε εδώ το πώς θα μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας και να δούμε. Έτσι, ελπίζω, έτσι εύχομαι και να δούμε τι θα γίνει με το άρθρο 6 που μιλά για την υπεράσπιση. Ελπίζω και να είναι εύστοχη η λύση και επομένω κλασικά σε αυτές τις διαπραγματεύσεις θα δούμε αν θα επιδειχθεί κάποια ευελιξία αλλά και το άρθρο 2 είναι ένα θέμα. Και ελπίζω όλα αυτά να έχουν ολοκληρωθεί αισίως μέχρι τα τέλη του έτους. Είναι η πρώτη φορά που σε ευρωπαϊκό νομοθετικό επίπεδο έχουμε ένα τέτοιο νομοθέτημα για τους ε, ανηλίκους. Και γι' αυτό λοιπόν και υπάρχουν πολλές προσδοκίες από πολλές χώρες. Πασχίζουμε λοιπόν προς αυτή την κατάσταση στις 12 του μηνός υπάρχει τριμερή συνάντηση, αλλά και άλλη στις 25 Νοεμβρίου ή στο Στρασβούργο. Και ενδιάμεσα πολλές τεχνικές συνεδριάσεις, οπότε υποφαινόμενοι και οι σκιώδεις προσπαθούμε ούτως ώστε να υπάρξει αίσιο Τέλος. Δεν είμαστε πολύ παρόντες τώρα, αλλά αν θέλετε να στείλουμε ένα μέλος της Επιτροπής να μάθει τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης γιατί είναι αρκετά σημαντικό το θέμα. Να στείλουμε λοιπόν τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ. Το επόμενο σημείο είναι η παρουσίαση της έκθεσης για την εφαρμογή το 14 του προγράμματος Περικλής για τις απομιμήσεις. Από το 12 είχε αρχίσει, όχι, είναι πρόγραμμα δράσης για την προστασία του ευρώ κατά των παραχαρακτών. Το κανονισμός 331 του 2014 το θέσπισε. Το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού αυτού λέει ότι πρέπει κάθε χρόνο να ενημερώνετε τακτικά, να πληροφορούμαστε. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν και μετά στους βουλευτάς, τους δύο παρόντες δηλαδή. Ορίστε Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μας δίνεται εδώ τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα αυτό. Να σας πω μερικά γενικά. Θα σας αναφέρω τις σημαντικότερες δράσεις που έγιναν να το 2014. Πριν όμως νομίζω ότι είναι σημαντικό να σας δώσω και μερικά στοιχεία για τις επαπειλούμενες παραχαράξεις και του ευρώ. Περίοδος 12 με 15 παρουσίασε μεγάλη παραχάραξη χαρτονομισμάτων ευρώ. Ας πούμε. Στα ετήσια στοιχεία της ΕΚΤ τον περασμένο Ιούλιο φάνηκε ότι το πρώτο ίμιση του 2015 450.000 παραχαραγμένα χαρτονομίσματα παρατηρήθηκαν, αύξηση δηλαδή 37% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμεινο του 2015. Υπάρχουν λοιπόν περισσότερα παραχαραγμένα ευρωχαρτονομίσματα. Τώρα για τα παραχαραγμένα νομίσματα, μεταλλικά νομίσματα και αυτά αυξάνονται. Στο Πόρτο Μαρίνο κοντά στην Νάπολη ας πούμε, θα τέλη του 14, 300.000 τέτοια νομίσματα, κέρματα ε, βρέθηκαν και είχαν παραχαραχθεί στην Κίνα. Τρίτον, αυξάνεται η ποιότητα των παραχαραγμένων κερμάτων ιδίως. Μοιάζουν πάρα πολύ με τα γνήσια και άρα είναι πολύ δύσκολο να τα βρουν μηχανές που δέχονται κέρματα, κερματοδέκτε. Όσο για τα στοιχεία που εγγυώνται την ασφάλεια των χαρτονομισμάτων όπως τα ολογράμματα, είναι πολύ εύκολο να πουληθούν διεθνώς για πολύ χαμηλές μάλιστα τιμές. Και αυτά τα χρησιμοποιούν βέβαια οι ομάδες οργανωμένου εγκουλήματος. Τα δεδομένα της Ιντερπόλ για το 2014 δείχνουν ότι 1,2 δισεκατομμύρια χαρτονομίσματα κατασχέθηκαν. με αξία 66 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, οι εκθέσεις της Ευρωπόλ δείχνουν ότι επειδή το ευρώ είναι το πιο κυκλοφορούν διεθνώς ε, νόμισμα και είναι και τόσο σταθερό, γίνεται πιο πολύ ελκυστικό για το οργανωμένο έγκλημα και άρα έχει συμφέρον να το παραχαράξει και να τα χρησιμοποιήσει τα παραχαραγμένα για ξέπλυμα βρωμίκου χρήματος. Αυτή η απειλή λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα σαν τον Περικλή που να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή. Πέρα από αυτά όμως θα ήθελα να αναφερθώ και στην οδηγία που εγκρίθηκε από τους συνομοθέτας και συζητήθηκε και στην Επιτροπή ΕΛΕΦ την 2014-62 που εγκρίθηκε όπως λέει το όνομά της το 14 και ε, χορηγεί αυξημένη προστασία κατά της παραχάραξης ευρώ. Να, εδώ λιγάκι τα γενικά στοιχεία της απειλής που αντιμετωπίζουμε. Τώρα για το πρόγραμμα Περικλής. Είναι βασικά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής πληροφοριών που είχε αρχίσει πριν από μερικά χρόνια αλλά επεκτάθηκε, παρατάθηκε. Μέχρι το 20. Καλύπτει δηλαδή 7 χρόνια και από το 13 και μετά. Αλλά δυστυχώς μόνο το 15 επεκτάθηκε και στις χώρες μέλη εκτός Ευρωζώνης. Γι' αυτόν τον λόγο το 2014 μόνο οι χώρες της Ευρωζώνης μπόρεσαν να υποφεληθούν από τον Περικλή. Εδώ μιλάμε για ένα ποσό περιορισμένο αλλά σημαντικό. 7,3 εκατομμύρια για τα 7 χρόνια λειτουργίας του. μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 20 δηλαδή. Το πράγμα αυτό έχει εξυγχρονιστεί σε σύγκριση με τον προκάτοχο του, έχει απλοποιηθεί και συμπεριλαμβάνει περισσότερες δραστηριότητες. Και η αξιολόγηση, επιτήρηση, εποπτεία του επίσης έχει αυξηθεί, δηλαδή τώρα πιο τακτικά πρέπει να δίνονται πληροφορίες για τα επιτρέχματα του περικλέους και αυτό βρίσκουμε ότι τώρα πληρούμε τις συνθήκες του άρθρου 20 που αναφέρατε κι εσείς και παρουσιάζουμε την έκθεση για το 14. Για το 14 λοιπόν ο προϋπολογισμός που χορηγήθηκε στον Περικλή ήταν 924.000 ευρώ και το μεγαλύτερο τμήμα του ποσού αυτού έχει χρησιμοποιηθεί. 10 σχέδια χρηματοδοτήθηκαν, 6 από τις αρμόδιες αρχές τριών χωρών της Ευρωζώνης, Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία. Και αυτό νομίζω οφείλεται στο ότι στις χώρες αυτές υπάρχουν οι, οι περισσότερες παραχαράξεις και γι' αυτό χρησιμοποιούν περισσότερο τον περικλή. Τέσσερα προγράμματα επίσης ανελήφθησαν από την Κομισιόν και τα δέκα αυτά μπορείτε να τα δείτε στην προσθήκη 1, το παράρτημα 1 της έκθεσής μας. Τα προγράμματα ήταν σεμινάρια, τεχνική εκπαίδευση, ανταλλαγές προσωπικού και μελέτες. Και ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές ολόκληρο τον κόσμο. Ιδιαίτερα το 14. Η Λατινική Αμερική, ας πούμε στη Χιλή, στην Κολομβία, έγινε ένα σεμινάριο για το ευρώ και το δολάριο και την παραχάραξη αυτών και στην Αλβανία και Τουρκία. Υπολογίζονται 662 εμπειρογνώμονες ότι συμμετέσχουν σε αυτά τα σεμινάρια που προέρχονταν και, από, και εκτός και εντός της Ένωσης. Οι περισσότεροι βέβαια από τις ευρωπαϊκές χώρες. Το επαγγελματικό τους ε, παρελθόν ήταν από την αστυνομία κυρίως, αλλά μεγάλη αριθμή και άλλων οργάνων από διαφορετικό παρελθόν. Προσωπικά κεντρικών τραπεζών, δικαστηρίων, Γενικά λοιπόν για να συνοψίσω το 14 συμμετέσχουν περισσότεροι εισαγγελείς και δικαστέ στον Περικλή. Έχει ένα πολύ ισχυρό στοιχείο περιφερειακής συνεργασίας και μπορεί να εκπαιδεύσει αστυνομικούς στην Κολομβία ας πούμε πράγμα που είναι πολύ σημαντικό παράδειγμα διότι υπάρχουν και στην Κολομβία κάτι hot spots που παράγουν παραχαραγμένα ευρώ και δαλάρια. σε συνεργασία πολλές φορές και με τις μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Παλιτιών. Υπάρχει διαφοροποίηση των προγραμμάτων τώρα και μελετών όπως την εξέταση του παρελθόντος των παραχαρακτών αλλά και μελέτες για τη βελτίωση της ασφάλειας των μελλοντικών κερμάτων γιατί πρέπει να σκεφτούμε και τη νέα γενεά των ευρωκερμάτων. Έγινε μια σημαντική διάσκεψη στη Φραγκφούρτη νωρίς το 2015 και που συνοργανώθηκε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπόλ όπου συνήλθαν 170 εμπειρογνώμονες από 40 έθνη και αυτό δείχνει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση του διεθνούς φαινομένου της παραχάραξης με σημαντικούς εταίρους όπως την Κίνα, η οποία βέβαια ακόμα δεν έχει εγκρίνει την συνθήκη της Γενέβης του 99, ε, του για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παραχαράξεως. χώρες πρέπει να προστατεύουν και το εθνικό τους νόμισμα και τα ξένα. Και τα ξένα. Έτσι το 2015 με την εφαρμογή του προγράμματός μας, του ετήσιου, συζητήσαμε τις νέες προτεραιότητες μαζί με τις χώρες μέλη, την ΕΚΤ και την Ευρωπόλ στα πλαίσια ενός προγράμματος εμπειρογνωμόνων της Κομισιόν. Και επίσης ταυτίστηκαν οι κύριες προτεραιότητες μας για φέτος ανά χώρα. Έχουμε ακόμη ως προτεραιότητα τον, την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και θα συνεχίσουμε φυσικά τις δραστηριότητες για την προστασία του ευρώ και σε τρίτες χώρες όπως τη Λατινική Αμερική. Η Επιτροπή επιτηρεί ακόμα την εφαρμογή του φετινού προγράμματος και μόλις έχουμε τα στοιχεία θα σας τα υπαβάλουμε και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Καταλήγω. Το πρόγραμμα Περικλής μέχρι το 20 συνεχίζει να είναι αποτελεσματικό και σημαντικό εργαλείο για την πρόληψη και καταπολέμηση της παραχαράξεως. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δύο είναι συνάδελφοι στην αίθουσα που θέλουν να ε, μιλήσουν η κυρία Τζινίτση και ο κύριος Αγγελάρ ενδεχομένως θα θέλατε να πείτε εσείς κάτι. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση και πολλά τα δεδομένα. Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επιτροπή, λέει η κυρία Κινίτση, για την έκθεση. Είναι το θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον και ελπίζω ότι και εγώ θα μπορέσω να συμβάλλω ενδιαφέρον και σημαντικό το θέμα τι να κάνουμε, θέμα είναι τέτοιο που θα ήθελε τριπλάσιο χρόνο. Μας απασχολεί σίγουρα πάντως. Είναι κάτι το οποίο καλύπτει πολλές διαφορετικές πτυχές. Πρώτα πρώτα είναι το θέμα και τεχνικό αλλά και νομικό. Είναι και κάτι που έχει να κάνει και με την έρευνα πάντως. Γιατί για άλλη μια φορά εδώ είναι ζήτημα συνεργασίας περισσότερων χωρών. Και όχι μόνο κρατών μελών. Όπως ακούστηκε, πρόκειται και για άλλες χώρες. Εκεί όπου σοβεί η παραχαράκηση και η βιβλία. Άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα τα ζητήματα, τα επιμέρους που ανακύπτουν, ακόμα και τα πιο δύσκολα. Τα σχετικά λοιπόν με ναι. Τι απειλέ αυτέ για το ευρώ και τώρα. Θα πρέπει να δούμε κάτι συγκεκριμένο ε, και για τα χαρτονομίσματα. Και αυτό πάντως το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε συνεργασία των διοικητικών αργών. Κυρίω όσον αφορά τις ερευνητικέ δραστηριότητε, Αλλά να έχουμε και δικαστική συνεργασία. Όχι μόνο συνεργασία με την Europol, και την Eurojust να υπάρξει συνεργασία και των επιμέρους χωρών. Αυτά τα ορίζει και τα προβλέπει το περικλής. Αλλά εμείς να προτείνουμε κάτι συγκεκριμένο. Ας πούμε, ειδική εκπαίδευση σε όσους αστυνομικούς ασχολούνται με αυτό το θέμα. Και πέραν από την αστυνομία και τους δικαστικούς να εκπαιδεύσουμε γιατί εδώ έχουμε θέμα πολύ ιδιόρυθμο. Αυξάνεται η η κυβήλια. Θα πρέπει ο μέρος να είναι αντίστοιχη και, και εντατική η συνεργασία μας ακριβώς όπως κάνουμε και για άλλους τομείς. Άρα, συνεργασία και στις έρευνες και στις καθαρά δικαστικές δραστηριότητες και με τις χώρες μέλη και με τρίτες χώρες και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, έχω, έχετε ήδη πάρει πολλές ερωτήσεις στην κυρία Συνήθεια. Σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Νομίζω ε, ότι πραγματικά χαίρομαι που αναφέρατε αυτά τα σημεία την δικαστική συνεργασία. Ακριβώς γι' αυτό οι δράσεις του Περικλή στην ουσία όλο και περισσότερο επικεντρώνονται στην δικαστική συνεργασία, στη δικαστική συνδρομή, την ανταλλαγή προσωπικού αλλά και πρακτικά εργαστήρια για τη συνεργασία στα οποία εκπροσωπούνται και συμμετέχουν οι δικαστικές αρχές. Για παράδειγμα έγινε στη Φραγκφούρτη τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έγινε μια τέτοια συνάντηση με εκπροσώπους από τις εισαγγελίε και τις δικαστικές αρχές οι οποίες συμμετείχαν, ήταν παρούσες, ε, όχι μόνο από κράτη-μέλη, αλλά και από άλλες χώρες όπως το Περού και η Κολομβία. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η συνεργασία να βελτιωθεί σε δικαστικό επίπεδο δεδομένες στις διεθνούς διάστασης που σας ανέφερα. Για την αστυνομική συνεργασία χαιρόμαστε ιδιαίτερα που για παράδειγμα οι Ιταλοί καραμπινιέροι έκαναν διαφορετικές, διάφορες ανταλλαγές προσωπικού με τις αντίστοιχες αρχές στην Αλβανία, τα Δυτικά Βαλκάνια και άλλες παρόμοιες περιοχές για να υπάρξει πρακτική εξάσκηση σε τεχνικό και τακτικό επίπεδο. Τα εθνικά κεντρικά επίσης γραφεία πρέπει να εγκατασταθούν σε κάθε κράτος μέλος και βάσει της συνθήκης της Γενέβης σε κάθε κράτος του κόσμου που έχει συνυπογράψει τη σύμβαση για να μπορέσει να υπάρχει συντονισμός στο θέμα της παραχάραξης και διεθνή συνεργασία. Αυτό είναι λοιπόν μια από τις προτεραιότητες του Περικλή και χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατή δράση για να βελτιώσουμε το επίπεδο των ερευνών σε τακτικό και νομικό επίπεδο φυσικά. Ευχαριστούμε τον κύριο Νόμου. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι μια διαδικασία σπάνια για την Επιτροπή μας, αν κατάλαβα καλά. Ο κύριος Τζαμπάνσκι κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο ερωτήματα. Το ένα ήταν το ερώτημα της 28 ε, Ιουνίου και το άλλο της Δευτέρας Ιουλίου του 2015 ως τώρα δεν έχουμε λάβει απάντηση από την ε, Επιτροπή. Ο κύριος Ζομπάνσκι δεν μπόρεσε σήμερα να έρθει εδώ για να γίνει η συζήτηση και γι' αυτό το λόγο δίνω το λόγο στην Επιτροπή για να μας εξηγήσει ακριβώς περί τίνος πρόκειται και ποια ήταν η διαδικασία και γιατί ο κύριος Τζαμπάνσκι δεν πήρε απάντηση. Ποιος θα μιλήσει εκ μέρους της Επιτροπής? Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα απαντήσω εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι σύμφωνα με τα δικά μας στοιχεία, οι έγγραφες απαντήσεις και σε αυτά τα δύο ερωτήματα έχουν ήδη αποσταλεί. Όσον αφορά στο ερώτημα 10.664, ε, η απάντηση στάλει στις 22 Οκτωβρίου και για την 1971 στις 21 Οκτωβρίου. Για την πρώτη ερώτηση, που η απάντησή της ε, εστάλει στις 2 Οκτωβρίου, η Κομισιόν θέλει να πει ότι τα ερωτήματα που καταθέτουν οι αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, που καταθέτουν οι κύριοι βουλευτές, βασίζονται σε μία συνέντευξη που έδωσε ο Ιταλός Πρωθυπουργός πριν γίνει η πολιτική συμφωνία για τη μετεγκατάσταση δεδομένου ότι πίστευε πως ε, δεν θα ε, λάβει το Συμβούλιο απόφαση βάσει των, αποφάσ... των προτάσεων της Κομισιόν για 40.000 και 20.000 άτομα αντίστοιχα. Στο μεταξύ όμως βρέθηκε η πολιτική συμφωνία για τους 40.000 τον Ιούλιο και η απόφαση εγκρίθη επισήμως ε, το Σεπτέμβρη. Επίσης, στις 22 Σεπτεμβρίου είχαμε επίσημη απόφαση και για την μετεκατάσταση 120.000 ανθρώπων. Άρα δεν νομίζω ότι η Επιτροπή χρειάζεται να πει κάτι παραπάνω. Γιατί στην ουσία θα μιλάμε έτσι με υποθέσεις για, θέματα τα οποία, για μέτρα τα οποία οι Ιταλοί θα έπρεπε να λάβουν βάσει των αποφάσεων που δεν θα είχαν ληφθεί. Θέλετε να πάω τώρα απευθείας στη δεύτερη ερώτηση. Ναι. ναι. Ωραία. Για τη δεύτερη ερώτηση, η οποία σχετίζεται με την κατάσταση στη Βουλγαρία και ο αξιότιμος κύριος βουλευτής ζήτησε η Βουλγαρία να έχει την ίδια αντιμετώπιση με την Ελλάδα και την Ιταλία όσον αφορά στις προτάσεις κατάσταση της Επιτροπής. Ένα από τα ζητήματα λοιπόν είναι ε, της απάντησης ε, είναι ότι η κατάσταση στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή δεν είναι το ίδιο με την κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ιταλία, ειδικά όσον αφορά τους άτυπους μετανάστες. Και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε για την άτυπη μετανάστευση στην Βουλγαρία, μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου φέτος είχαμε 26.000 άτομα που έφτασαν παράνομα και θέλησαν να περάσουν από τα σύνορα της χώρας. Φυσικά τα νούμερα για την Ιταλία και την Ελλάδα είναι πολύ διαφορετικά. Δεν έχουμε ακριβώς συγκρίσιμα στοιχεία για όλη την περίοδο, αλλά για την Ελλάδα είναι πάνω από τα 30.000 τα άτομα, ενώ για την Ιταλία είναι 140.000. Αλλά φυσικά η Κομισιόν συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση στη Βουλγαρία και σε όλα τα κράτη-μέλη στενά. Και είναι έτοιμη όποτε χρειαστεί να προτείνει παρόμοια μέτρα μετακατάστασης, ειδικά αν υπάρξει μια έκτακτη ανάγκη όπως αυτή που είχαμε σε αυτά τα άλλα δύο κράτη-μέλη. Thank you. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Δεν είναι εδώ ο κύριος Ζαμπάσκη, αλλά είναι η βοηθός του εδώ. Μα αν θέλετε μπορείτε να σημειώσετε. Εδώ εξαντλήθηκε η μερίσια διάταξη. Η προσεχή συνεδρίαση 16 Νοεμβρίου. Καλησπέρα. Thank you.